Ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην ακρόαση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Σας καλωσορίζω από πλευράς της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, Οπότε απευθείας να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σέρτζο Γκαϊτάνο Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω τους προσκαλεσμένους μας και ακριβώς για να μην χάνουμε χρόνο θα ήθελα να πω ότι στην Επιτροπή μας εδώ και λίγο χρόνο έχουμε αρχίσει μία συζήτηση επί της οδηγίας που αποτελεί αντικείμενο της σημερινής ακρόασης. Θα έπρεπε η οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων να αναδειχθεί ως μοντέλο διακυβέρνησης της ευρωπαϊκής επιχείρησης. Τουλάχιστον αυτό ευχόμαστε. Ξέρετε ότι έχουμε προσδώσει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα και μας απασχολεί από το 1993 από τη Λευκή Βίβλο του Ζακ Delors όπου η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων η κοινωνική εταιρική ευθύνη μας απασχόλησε και νομίζω ότι όλοι το συμμεριζόμαστε αυτό. Διανύσαμε πολύ δρόμο, ασχοληθήκαμε με θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υπάρχουν και συναφή κεφάλαια όπως αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα το απόγευμα το πνεύμα της οδηγίας ή καλύτερα της πρότασης της Επιτροπής είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνους. Υπάρχουν όμως στοιχεία που νομίζω ότι δεν συμμεριζόμαστε ούτε εμείς ούτε άλλοι συναδελφοί. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν και να επανεξεταστούν βασικός στόχος είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους μετόχους και διευκόλυνση διαβίβασης δεδομένων σε όλη την αλυσίδα ενδιάμεσων και να μας απασχολήσει και το θέμα της ψήφου των μετόχων. Σύμφωνα με τις ε, αρμοδιότητες τους, Ξέρετε ότι πολλοί από τους μέτοχους δεν ορίζονται επαρκώς, διότι ο βασικός πυρήνας των μετόχων αποτελεί ε, μετόχους μειοψηφίας. Το θέμα της διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό, το έχω πει πολλές φορές και αυτός είναι και ο απότερος στόχος των εργασιών μας. Αυτό αφορά τους θεσμικούς επενδυτές και το, το βασικό πυρήνα των διαχειριστών και των ε, κατεξουσιοδότηση συμβούλων. Το θέμα των διαχειριστών και των διευθυντών είναι ύψης της σημασίας και πάνω απ' όλα οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να επιλέγουν βραχυπρόθεσμους στόχους. Και ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει διαφάνεια, αντιμετωπίζουμε φαινόμενα ιδιαίτερα επώδυνα για επιχειρήσεις, δηλαδή χάνεται η αξιοπιστία τους. Πρόκειται για επιχειρήσεις ε, που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση και όπου ε, πρόσφεραν πολύ ψηλέ αμοιβέ ε, στα διευθυντικά στελέχη και στη συνέχεια είχαν και προβλήματα ρευστότητας. Το θέμα λοιπόν της αμοιβή θα πρέπει να το δούμε και στα πλαίσια της συμπληρωματικής αμοιβή ή των ε, συμπληρωματικών αμοιβών. Υπάρχουν δηλαδή πριν και benefits τα οποία δεν είναι ανάλογα με τους στόχους της επιχείρησης, είναι ιδιαίτερα δυσανάλογα μέσα στα πλαίσια της ε, πρακτικής διαχείρισης της επιχείρησης. Επίσης, η έλλειψη διαφάνειας και ελέγχων οδήγησαν σε αρνητικά σχήματα, διότι τα θέματα της αμοιβή και των αμοιβών είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν. Αυτό θα το ε, δούμε και σήμερα το απόγευμα στις συζητήσεις, ξεκινώντας από αυτά τα σημαντικά ζητήματα που είναι ύψης σημασίας. Ξέρω ότι υπήρξαν σχόλια στα, στις άτυπες ε, ανταλλαγές απόψεων μεταξύ ημών και γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο πρώτο αυτό τμήμα ή μέρος της συζήτησης. Θα θέλαμε βεβαίως να μας πείτε και τη δική σας κρίση, τα σχόλιά σας, έτσι ώστε η οδηγία αυτή να αποτελέσει έναυσμα της επανεκκίνησης της εταιρικής διακυβέρνησης. Δηλαδή αφορά όχι μόνο τους μετόχους αλλά και τους εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους φορείς. Για να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία. Βεβαίως έχει σημασία η διαφάνεια και η συνοχή, ιδιαίτερα σε όσον αφορά τις δραστηριότητες της επιχείρησης όπως το καθεστώς αμοιβών και ευθυνών καθώς και δικαιωμάτων, καθώς και μία διάκριση μεταξύ, μεταξύ ε, δραστηριοτήτων και συναλλογών. Να μην υπάρχει λοιπόν κερδοσκοπία, η οποία δεν σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα σταματήσω εδώ. Ήθελα απλώς να αναφερθώ σε ορισμένα σημαντικά σημεία που θα μας απασχολήσουν και μετά θα τα δούμε εν λεπτομερία. Θα σας ακούσω με μεγάλη προσοχή. Και στο τέλος της συνεδρίας αυτής θα προσθέσω ορισμένα σχόλια, καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πέντε διακεκριμένους ομιλητές σήμερα το απόγευμα τους οποίους καλωσορίζω θερμότατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί φίλοι, βεβαίως ε, είστε εξέχοντες εμπειρογνώμονες, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να τηρήσετε το χρόνο σας. Δυστυχώς ε, ο καθένας θα έχει μόνο 10 λεπτά. Λοιπόν, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ όσο πιο βιανικά μπορώ να τηρήσετε το χρόνο σας. Πρώτος ομιλητής είναι η Carrie Waring, ε, επικεφαλής ε, της οργάνωσης ICGN. Έχει το λόγο. Καλό σας απόγευμα. Είμαι η Κάρι Βέρινγκ, διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Δικτύου Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο George Ντάλλας ε, βρίσκεται εδώ κοντά. Σας ε, ευχαριστώ, είμαι ευγνώμων γιατί μπορώ να σας ε, μιλήσω για την αναθεώρηση της οδηγίας των δικαιωμάτων μετόχων. Το δίκτυο συστάθηκε 20 χρόνια πριν και βασίζομαι στην προώθηση των δικαιωμάτων των μετόχων. Έχουμε 160, 650 συγγνώμη, μέλη σε 50 χώρες και ασχολούμαστε με την διαχείριση στοιχείων ενεργητικού που υπερβαίνουν τα 18-3 δολάρια. Τα σχόλιά μου λοιπόν θα σχετίζονται με, αυτή την, ε, ε, με αυτό το θέμα ευρεία ευέλεια. Μας ενδιαφέρει λοιπόν αυτό το θέμα που σχετίζεται και με τα δικαιώματα ψήφου. Επίσης, συμφωνούμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη δέσμευση μεταξύ επιχειρήσεων και επενδυτών, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και οικονομία. Για τους λόγους αυτούς θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στα εξής. Καταρχήν θα ήθελα να δούμε την ε, διακυβέρνηση αυτή μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της κεφαλαίου αγοράς. Δεύτερον, θα ασχοληθώ με συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με τις ε, δεσμεύσεις των μετόχων και την ευθυγράμμισή τους. Τρίτον, θα ασχοληθώ με το θέμα της αμοιβή και της ε, ψηφοφορίας, της διασυνοριακής ψηφοφορίας. Η διακυβέρνηση αυτή έχει μεγάλη σημασία γιατί θεωρούμε ότι η χρηστή διακυβέρνηση σχετίζεται με την διαχείριση του κινδύνου μέσα στα πλαίσια της εποπτείας και της ρύθμισης. Έτσι, δεν χρειάζεται να προβούμε σε αποσβηστικές ρυθμίσεις. Η καλή εποπτεία της χρηστής διαχείρισης σχετίζεται με τα δικαιώματα των ε, μετόχων και της διαφάνειας μέσα στα πλαίσια της άσκησης των δικαιωμάτων τους, μέσα στα πλαίσια της σωστής πληροφόρησης. Εάν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, σε αυτή την περίπτωση μπορούν να θεωρήσουν τις επιχειρήσεις υπόλογες και να διαχειριστούν τους κινδύνους θεωρούμε ότι έχει μεγάλη σημασία να χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο της κυριότητας μετοχών και έτσι το δίκτυο μπορεί να βοηθήσει τους μετόχους να ασκήσουν τις ευθύνες και τις, τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά τους. Σε σχέση με τη δέσμευση των μετόχων θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, δημοσιοποιήσουν τα σχέδια αυτά όμως, μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων, συγκεκριμένες εμπειρίες θεωρούμε ότι το άρθρο αυτό δεν καθιστά σαφές πώς τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και σε τι χρονικό πλαίσιο. Οι αρχές παγκόσμιας διακυβέρνησης του δικτύου σχετίζονται με τους επενδυτές και τα στοιχεία που θα πρέπει να κοινοποιήσουν στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να κινηθούμε πέρα από τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες και να κινηθούμε και σε δεοντολογικά και κοινωνικά ζητήματα. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους εθνικούς κώδικες δεοντολογίας των επενδυτών που βασίζονται στις αρχές του δικτύου. Και πολλά μέλη του δικτύου μας προβαίνουν σε δηλώσεις στην ιστοσελίδα τους. Επίσης, έχει σημασία να λάβουμε υπόψη ότι οι εταιρείες χαρτοφυλακίου θα πρέπει να λάβουν υπόψη συγκεκριμένες προτεραιότητες με βάση την φύση της εντολής ή το μέγεθος των εταιριών χαρτοφυλακίου μέσα στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής. Σε σχέση με τη συλλογική δέσμευση θεωρούμε ότι σε περιπτώσεις εξαγοράς δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές και οι μέτοχοι δεν θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες, διότι πολλές φορές έρχονται σε επαφή με συναδέλφους μέσα στα πλαίσια της διασυνοριακής συνεργασίας, έτσι ώστε να βελτιώσουν την εταιρική διακυβέρνηση. Επίσης, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Το δίκτυο πολλά χρόνια, για πολλά χρόνια θεώρησε ότι οι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να αναγνωρίσουν αυτή την ευθύνη τους μέσα στα πλαίσια των δικαιωμάτων των τελικών δικαιούχων. Και αυτό αφορά και τους συμβατικούς όρους που διέπουν τη, τους θεσμικούς επενδυτές μέσα στα πλαίσια και της διαχείρισης ε, από πλευράς των διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν πάντα να δημοσιοποιούνται, διότι αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Γι' αυτό, για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι προσέγγιση θα πρέπει να προωθήσουν και επίσης αυτό αφορά και τους διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού. Προωθούμε τα δικαιώματα των μετόχων, ιδιαίτερα δυνάμει του άρθρου 9, μέσα στα πλαίσια των αμοιβών του διευθυντικού προσωπικού. Πολλές φορές οι μέτοχοι θεώρησαν ότι τα σχέδια αμοιβών θα πρέπει να εγκρίνονται από τους ίδιους πριν εφαρμοστούν. Οι μέτοχοι δεν μπορούν να διαδραματίσουν συγκεκριμένο ρόλο αν τα δικαιώματά τους είναι περιορισμένα και θα πρέπει να μπορούν να επηρεάζουν τα πράγματα ανάλογα με, το, ε, με τα κεφάλαια κινδύνου τα οποία επενδύουν. Και θεωρούμε ότι ο διάλογος δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιαστεί στις αμοιβέ κατά άλλων παραγόντων όπως η στρατηγική, ο κίνδυνος και η αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τα, τα δικαιώματα των ε, μετόχων και μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και η αρχή της πλήρεξουσιότητας ε, ή το ε, share blocking. Μέσα στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ισχύουν οι οδηγίες περισσότερο, για περισσότερο χρονικό διάστημα από το απόλυτα αναγκαίο και αναγνωρίζουμε την ανάγκη ευελιξία σε ορισμένες αγορές. Υποστηρίζουμε προτάσεις για την επιβεβαίωση ψήφου, διότι πολλές φορές οι επενδυτές δεν λαμβάνουν πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματός τους, έτσι ώστε να πούν στους δικαιούχους ότι η ψήφος τους ελήφθη υπόψη. Ως προς τις ταπάνες θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει προωθημένη διαφάνεια σε επίπεδο εισφορών, έτσι ώστε το, οι εμπλεκόμενες δαπάνες να είναι ανάλογες με, τους, ε, ε, με τα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης έχω παρουσιάσει ένα γραπτό έγγραφο σε σχέση με την αναθεωρημένη ε, οδηγία, το οποίο έχω δώσει στην κριτική επιτροπή. Ο Νίλς Λέμονς είναι επίσης εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να μας υποβάλλετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο δεύτερος ομιλητής, η δεύτερη ομιλήτρια, είναι η κυρία Σουζάνα Χάν, Γενική Γραμματέας ε, των Ευρωπαίων Εκδοτών Μετοχών. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ του Ευρωπαίου Εκδότε, European Issuers. Ε, είμαστε μια πανευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εισηγμένων εταιριών ε, στην Ευρώπη στα μέλη μας περιλαμβάνονται και εθνικές ε, ενώσεις και μεμονωμένες εταιρείες. Στόχος μας είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορεί οι εταιρείε να συγκεντρώνουν κεφάλαια μέσω των δημόσιων αγορών και να έχουν σε αποτέλεσμα την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Άρα θέλουμε κεφάλαια αγορέ να υπηρετούν τα συμφέροντα των τελικών χρηστών και των εκδοτών και των επενδυτών δηλαδή, μεταξύ άλλων. Πριν ξεκινήσω να σας ε, εκθέτω τις μεμονωμένες προτάσεις της θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για το ρυθμιστικό και το οικονομικό πλαίσιο εντό ε, του οποίου προτείνεται η εν λόγω οδηγία. Τα τελευταία δέκα χρόνια περίπου Υπήρξε πολλέ ρυθμίσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για τι μη χρηματοπιστωτικέ εταιρείε. Αρχικά το σχέδιο δράση για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, το σχέδιο δράση για την εταιρική σχέση και το ε, διακυβέρνηση και το εταιρικό δίκαιο και με την χρηματοοικονομική κρίση στη συνέχεια επηρεάστηκαν και οι ε, εταιρείε από του χρηματοπιστωτικού αυτού κανόνε. Κάτι το οποίο όμως ε, έλειπε ήταν η αναθεώρηση της υλοποίησης ε, της οδηγίας για τα Δημήτρα των μετόχων από το 2007 ή τέλος πάντων δεν μελετήθηκε το σωρευτικό αποτέλεσμα όλων αυτών των ρυθμίσεων που προανέφερα. Ε, τι, πώς επηρέασε όλη αυτή η τελος παντων δεν μελετηθηκε το σορευτικο αποτελεσμα ολων αυτων των ρυθμισεων που προανεφερα τι πως επηρεασε ολη αυτη η ρυθμιση και για το ρόλο παραδείγματος χάρη των ανεξάρτητων διευθυντών. Ουσιαστικά έγιναν μεν διαβουλεύσει, αλλά δεν έγιναν πραγματική ανάλυση των επιλογών και των πιθανών λύσεων. Άρα η πρόταση δεν έχει τη στήριξη των εταιριών σε πολλές λεπτομέρειες, διότι θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, οι ρυθμίσεις δεν είναι σχεδιασμένοι κατά ανάγκη ε, κατάλληλα για τις επιχειρήσεις, ούτε προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσει. Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ανάπτυξη και επασχόληση, άρα χρειάζεται εταιρείε που μπορούν να παράγουν κέρδο και να απασχολούν περισσότερου εργαζομένου. Αυτό το οποίο θα ήθελαν λοιπόν οι εταιρείε είναι ένα πιο σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσει εργασία όταν εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Πρόσφατα εξετάσαμε το ζήτημα του ρόλου των εισημένων εταιριών. Έχουμε μάλιστα δημιουργήσει και μια ειδική ομάδα, ένα task, μια task force στι ΗΠΑ. Αυτό έγινε πριν από λίγα χρόνια και είδαμε ότι διπλασιάζονται τα ποσοστά απασχόληση των εταιριών αφού εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Αυτή είναι η τάση. Παρατηρήσαμε επίσης ότι υπάρχουν εισηγμένες εταιρείε ε, αρκετές, αλλά μειώνεται ο αριθμός τα τελευταία 15 χρόνια. Μπορεί να έχουν ένα διπλάσιο μέγεθο ε, ή να χρειάζεται να έχουν διπλάσιο μέγεθο όμω για να έχουν πρόσβαση πλέον ε, στι αγορέ οι εταιρείε σε σχέση με το τι τα πριν από 20 χρόνια. Βλέπουμε ότι φαίνεται να συνιστά μεγάλο άκτος για πολλές επιχειρήσεις, είτε τον εισαχνούν, το να παραμείνουν εισηγμένες ε, στο χρηματιστήριο, γι' αυτό στρέφονται σε άλλες σε άλλους, ε, άλλες μεθόδους. Και αυτό κυρίως οι μικρότερες εταιρείε. Έχουμε το κόστος και το διοικητικό κόστος και το διαχειριστικό διοικητικό κόστος για αυτές τις ε, επιχειρήσεις. Οπότε πολλές φορές αυτό αποτελεί αντικίνητρο για την εισαγωγή αυτών των επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο. Τι είδους αγορές λοιπόν θα θέλαμε που θέλουν, σε τι πλαίσιο θέλουν να κινούνται οι επιχειρήσει είναι αυτές οι οποίες στηρίζουν ε, την πολυμορφία των διαφόρων κωδικών εταιρική διακυβέρνησης. Έχουμε το ρόλο των ε, διοικητικών συμβουλίων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τη διαφοροποίηση, ανάλογα με τη χώρα και ούτω καθεξής. θέλουμε να υπάρχει μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ και μετόχων. Γι' αυτό στηρίζουμε τους στόχους της οδηγίας που θέλει να προωθήσει τη συμμετοχή, τη δέσμευση. Βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ε, ανάλογα με το κράτος μέλος για τον ρόλο που θα πρέπει και μπορούν να διαδραματίσουν οι μέτοχοι για τη στήριξη της εταιρική διακυβέρνησης και τι ρόλο έχουν οι μέτοχοι αφενός και το Διοικητικό Συμβούλιο αφετέρου. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, μπορεί να έχουν οι μέτοχοι ε, τους πόρους και τα μέσα για να αναλύουν τις προτάσεις και να τις ψηφίζουν. Ε, σε αυτή την οδηγία είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών πρόταση ψήφου ε, σε μετόχους για πολλές συναλλαγές. Εμείς όμως δεν είμαστε σίγουροι για το κατά πόσον είναι ενδεδειγμένο αυτό ή κατά πόσον η αναθεώρηση ή η επιβεβαίωση από τους ε, διευθυντές που δεν συμμετέχουν σε αυτή τη συναλλαγή, στη συναλλαγή αρκεί. Δηλαδή μπορούν οι μέτοχοι, έχουν το χρόνο, έχουν τα μέσα για να αναλύσουν όλες αυτές τις ε, προτάσεις. Μήπως αυτό οδηγήσει σε καθυστερήσεις στις συναλλαγές και μπουν έτσι σε μενεκτική θέση έναντι των ιδιωτών ανταγωνιστών αυτές τις σημαίνες εταιρείε. Και αν υπάρχει ψηφοφορία, μήπως αυτό θα μπορούσε να περιοριστεί σε σημαντικότερες συναλλαγές. Είναι μια άλλη απόρρια εφόσον αυτή τη στιγμή δεν προβλέπονται αποτελεσματικές εξαιρέσεις λόγω του ευρύτατου πεδίου. Ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις πιστεύουμε ότι θα πληγούν, θα πληγούν ε, έντονα 5% ε, με ανώτατο όριο 50 ε, εκατομμυρίων ευρώ είναι τελείως διαφορετικό από μια εταιρεία, από 5% μιας εταιρείας που έχει 5 δισεκατομμύρια ανώτατο όριο, market cap. Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, θα προτιμούσαμε αυτό να αφαιθεί στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, η ε, επιλογή ψήφου είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων, περιοριτική, δεσμευτική, αυτό να είναι εθνική αρμοδιότητα και να μην ορίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιο πολύ ε, να τονίζει τα ζητήματα της αποκάλυψης ε, των πληροφοριών το ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, έχουμε τους πληροεξούς συμβούλους που θα πρέπει να κάνουν την ανάλυση. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση γιατί η εταιρική μπορεί να μην είναι αποτελεσματικοί. Οι αναλυτές της εταιρικής διακυβέρνησης το 80% του χρόνου τους το δαπανούν στις αποδοχές, όπως το είδαμε σε μια συνεδρίαση της ε, Ιρλανδικής Προεδρίας πέρυσι, το είπε ένας επενδυτής. Άρα δεν έχουν πολύ χρόνο για οτιδήποτε άλλο. Τώρα, ε, δικαίωμα ψήφου, ένα για την έκθεση, ένα για την πολιτική. Αν αλλάξει όμως, ε, πουλήσουν κάποιες μετοχές, έρθουν άλλοι μέτοχοι στη θέση τους που έχουν άλλες απόψεις, ψηφίσουν διαφορετικά, η επιχείρηση πώς πρέπει να αντιδρά, πώς θα αντιμετωπίζει τέτοιου είδου αλλαγέ. Ό,τι αφορά τώρα την αναγνώριση ή ταυτοποίηση των μετόχων. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει η εταιρεία να έχει το δικαίωμα να αναζητά την αναγνώριση, την ταυτοποίηση των μετοχων πιστευουμε οτι θα πρεπει η εταιρεια να εχει το δικαιωμα να ζητα την αναγνωριση την ταυτοποιηση των μετοχων Θέλουμε να έχει το δικαίωμα η εταιρεία, δεν θέλουμε να, ε, αυτό που προτείνει η Κομισιόν για τους μεσάζοντες. Και δεν νομίζουμε επίση ότι θα πρέπει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν νέο μηχανισμό επειδή υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στην Ευρώπη. Η εταιρεία θα πρέπει να μπορεί να προσεγγίζει οποιονδήποτε στην ε, αλυσίδα. Και θα πρέπει η εταιρεία να έχει το δικαίωμα να επιλέξει το επίπεδο ταυτοποίηση, είτε στο επίπεδο του fund manager, είτε στο συνταξιδοτικό ταμείο, για παράδειγμα. Δεν είμαστε υπέρ αυτοεξαίρεση, δεν είμαστε υπέρ ενό κατοφλίου κάτω από το οποίο δεν θα μπορεί να υπάρχει αυτή η ταυτοποίηση. Επειδή έχουμε γενικά ε, διάχυτη ιδιοκτησία σε πολλέ μεγάλε εταιρείε. Και οι πολλοί, υπερβολικά πολλοί άριθμοι μέτοχοι θα εξαιρούνται σε μια τέτοια περίπτωση αν έχουμε μια εισηγμένη στο γερμανικό χρηματιστήριο DAX 30 εταιρεία που έχει 175.000 μετόχους, από αυτούς θα έπαιρνε κανείς λεπτομέρειες μόνο για 100 μετόχους. Τέλος, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον με βάση τη δική μας εμπειρία η εταιρεία θα πρέπει να ε, έχει ε, τα δικαιώματα, να δεκρατά τα δικαιώματα μερισμάτων και ψήφου. Είναι σημαντικό αυτό το σύστημα λοιπόν ταυτοποίησης για να μπορεί η εταιρεία να έχει επαφή με τους μετόχους, για να κατανοεί ποιες είναι οι προθέσεις πίσω από την ψήφο τους και ε, για τις διατάξεις που αφορούν τις αποδοχές και για τις ε, συλλαγές συνδεμένων μερών. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των μετόχων, θέλουμε και ε, είναι ο στόχος μας οι επενδυτές να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους, συζητούμε ε, στις συναντήσεις μας μετά την οδηγία του 2007. Θέλουμε αυτά τα επιχειρησιακά ε, πρότυπα και αρχές να λειτουργήσουν σωστά. Στηρίζουμε λοιπόν τη χρήση ε, των προτύπων που έχουμε, General Meeting Standards, αλλά το πρόβλημα πολλές φορές έχει να κάνει με την αλυσίδα των μεσαζόντων 28 μέρες ε, νωρίτερα ε, δημοσιεύονται κάποια έγγραφα, αλλά οι επενδυτές θα λαμβάνουν 7 ημέρες μόνο. Να, λοιπόν, να σταματήσω εδώ γιατί έχω υπερβεί ελαφρώς το χρόνο μου. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτος, τρίτη ομιλήτρια, η κυρία Άμπιγκελ Χάρον, που είναι επικεφαλής της ε, οργάνωσης Επενδυτές Αβίβα για υπεύθυνες επενδύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να δώσω την προπτική ενός επενδυτή και χαίρομαι που μπόρεσα να φύγω από το βροχερό Λονδίνο και να έρθω στις βροχερές Βρυξέλλες. Η Αβίβα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ε, συνταξιδοτικών κεφαλαίων και ασφαλίσεων. Έχουμε ενεργητικά ύψους 300 δις στο Ηνωμένο Βασίλειο την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Λιθουανία. Είμαι υπεύθυνη για τις ε, υπεύθυνε επενδύσεις. Είμαι λοιπόν υπεύθυνη για το επενδυτικό τμήμα. Συναντώμε λοιπόν με εταιρείε στις οποίες έχουμε επενδύσει για να δούμε πώς σέβονται θέματα, για παράδειγμα, φύλων και μειονοτήτων στα Δυτικά Συμβούλια, το ύψος ε, των αμοιβών, οικονομική ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή. Έχουμε λοιπόν μια στρατηγική δέσμευση για, υπεύθυνες, για υπεύθυνε επενδύσει και είμαι υπεύθυνη για το πώ ψηφίζουμε στι ε, Γενικέ Συνελεύσει Μετόχων. Ε, συναντιέμαι με εκπροσώπους τη ε, κοινωνία των πολιτών και άλλου επενδυτέ. Συμμετέχω λοιπόν πολύ σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση των κεφαλαίων αγορών και έχουμε μιλήσει γι' αυτό σε διάφορες εκδηλώσεις. Δεν είμαστε υπέρ της βραχυπρόθεσμης προοπτικής και χαιρόμεθα που η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η επίπτωση στην κλιματική αλλαγή είναι εντός των προτεραιοτήτων του Προέδρου Γιούγκερ. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ε, δέσμευση σε όλες τις χώρες. Κατά τη γνώμη μου, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να παίξουν ζωτικό ρόλο, νομοθετώντας και αξιοποιώντας και τις άλλες δυνατότητες που έχουν για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Καλωσορίζω λοιπόν τις ε, προσπάθειες του Προέδρου Γιούγκερ και των Επιτρόπων ε, Χιλ και Τίμερμαν για υπεύθυνη πολιτική επενδύσεων. Και χαιρετίζω και την πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση της Ευρώπης 2020. Εμείς θέλουμε να θεωρήσουν οι επόμενες γενιές ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διασφαλίσουμε το μέλλον τους. Έχω συμμετάσχει σε αυτό. Είχα μιλήσει γι' αυτό, για παράδειγμα, αρχές του χρόνου σε μια εκδήλωση για το θέμα αυτό στην Αθήνα. Είπα λοιπόν ότι πρέπει να αφήσουμε μια καλή κληρονομιά και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσης έχουν καλό ιστορικό νομοθετώντας από την οδηγία για τις εκθέσεις, για τις μη ε, χρηματοπιστωτικές απόψεις των επενδύσεων και για τις υπεύθυνε επενδύσεις. Γιατί νομίζουμε λοιπόν ότι είναι αναγκαία αυτή η οδηγία. Να είμαι σαφέστατη. Είμαστε απολύτως υπέρ αυτή τη οδηγία. Αντιμετωπίζει μια σειρά από ελλείψεις των αγορών και αποτυχίες των αγορών Πιστεύω ότι θα βελτιωθεί έτσι η εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές Κέφαλε αγορές και θα έχουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη. Κάτι άλλο. Το είπαμε ήδη. Μία από τις βασικές αιτίες της κρίσης του 2008 ήταν ότι το βραχυπρόθεσμο κέρδος ήταν προτεραιότητα. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει τι θα γίνει και πόσα θα κερδίσουμε το επόμενο τρίμηνο. Δεν βλέπαμε λοιπόν τις μακροπρόθεσμες ε, προβληματικές τάσεις. Αυτό εξακολουθεί να είναι αποτυχία των αγορών και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η ενημέρωση είναι η αρτηρία των κεφαλαίων αγορών, οι αρτηρίες. Και αν η ενημέρωση δίνεται μόνο για βραχυπρόθεσμα θέματα, τότε και η αποφάση για τις επενδύσεις και η κατάσταση των αγορών θα είναι βραχυπρόθεσμη, για αντιμετώπιση των αγορών, η προοπτική τους. Είναι λοιπόν ε, ζωτικό αυτό. Η μακροπρόθεσμη προοπτική και ενημέρωση. Δεν πρέπει να δυνατήσει. Αυτό πρώτα απ' όλα λοιπόν ενημέρωση για να μπορούμε να καθορίσουμε την ταυτότητα των μετόχων. Αυτό θα βοηθήσει να σταματήσουν μερικές από τις ε, αδυναμίες στην διατήρηση ε, των ε, επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν οι μέτοχοι να αξιοποιήσουν το βάρος τους για να βελτιωθεί η ε, εταιρική διακυβέρνηση. Και πρέπει επίσης να μπορούμε να βρούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν είναι συνεπής έναντι των υποχρεώσεων τους. Πρέπει περισσότερο και οι επενδυτές και οι διαχειριστές ενεργητικού να το λάβουν υπόψη αυτό. Φέτος, για παράδειγμα, επειδή παρενέβημεν σε μία ε, επενδυτική εταιρεία σταματήσαμε ε, κάποιες ε, κάποιες εξορίξεις σε ένα εθνικό πάρκο στο Κονγκό. Ζητήσαμε να υπάρξει μελέτη επιπτώσεων και βεβαίως στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα άλλο θέμα που πρόσφατα έχει αναφερθεί είναι πόσα λεφτά πήρε για να εισέλθει μια συγκεκριμένη εταιρεία σε ένα ε, επενδυτικό κλάδο. Βεβαίως, ε, επειδή είμαι υπεύθυνη για αυτό το τομέα, θα τα έλεγα αυτό, αυτά, αλλά κάνουμε όλο και περισσότερες προσπάθειες, ούτως ώστε να ε, είναι σαφές πώς έχουν ψηφίσει οι ΜΕΝ και οι ΔΕ για τα πιο δύσκολα θέματα και τα πιο δυσάρεστα θέματα στις γενικές συνελεύσεις και πρέπει να ξέρουν όλοι πώς ψηφίζουν οι ε, μέτοχοι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια γενική συνέλευση όπου μελετήσαμε ε, κατά πόσον είναι υπεύθυνοι οι επενδυτές και όχι οι εταιρείες. Ήμουν εγώ και επικεφαλής των ε, επενδύσεων και είχαμε μια σειρά από μέλη διοικητικών συμβουλίων ε, συνταξιοδοτικών ταμείων και μας ρωτήσανε σε επίμαχα θέματα πώς ψηφίσαμε, τι κάναμε για να παρακολουθούμε πώς γίνονται οι επενδύσεις και που γίνονται, σε τι εταιρείε γίνονται. Έχουμε λοιπόν τέτοιου τύπου διάλογο με τους πελάτες μας. Τώρα, οι αμοιβέ των εκτελεστικών στελεχών. Πρέπει να, είναι, να υπάρχει διαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται. Πρέπει να συνδέεται με τη στρατηγική της επιχείρησης και πρέπει να συνδέεται και με μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική. Εάν δεν ε, διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο, τότε αξιοποιώ τις δυνατότητες που έχω να ψηφίσω, την εξοδότηση που έχω να ψηφίσω, για να καταψηφίσω τις αποφάσεις. Έτσι στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα. Βέβαια πολλά πρέπει να κάνουμε ακόμη, αλλά έχει υπάρξει πρόοδος, ιδιαίτερα σε αγορές όπου μπορούμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις των αμοιβών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα για το πώς ψηφίζουμε. Ταξί δύο. Πρώτον, θεωρούμε ότι οι πληρεξούσιοι σύμβουλοι είναι πολύ χρήσιμοι για να συλλέγουμε στοιχεία, γιατί ασχολούμεθα με 4.000 ε, επιχειρήσεις το χρόνο, είναι πολλή δουλειά. Και δεύτερον, είναι απογοητευτική η έλλειψη διαφάνειας. Δεν μπορώ καν να διαπιστώσω αν έχει ληφθεί υπόψη η ε, ψήφος, που, ε, η ψήφος μου, παρά το ότι έχω κάνει τόσες προσπάθειες για να μπορέσω να ψηφίσω. Θα ήταν πολύ εύκολο να ψηφίζω υπέρ των πάντων που προτείνονται. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχουν προτάσεις να είναι πιο εύκολο να δούμε ποιοι είναι οι ε, μέτοχοι σε πολυεθνικές εταιρείε και να είναι σαφές ότι έχουμε ψηφίσει σωστά με βάση τις ε, εντολές τους. Βεβαίως ε, δεν μας ικανοποιεί ότι μειώθηκε η αυστηρότητα των ε, μέτρων για τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. Αυτά τα δικαιώματα ε, υπάρχουν ήδη σε πολλές χώρες και δεν έχουν υπάρξει παρενέργειες. Εάν βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση, πιστεύω ότι θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη στις εταιρείε στις χώρες της Ένωσης, γιατί σε πολλές ε, χώρες της Ένωσης υπάρχει πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία. Κατά λίγο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και πλήρης λογοδοσία σε όλη την αλυσίδα μεταξύ των εταιριών και των τελικών επενδυτών. Και αυτή η οδηγία είναι σημαντικό βήμα σε αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό την υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα. Όσο περισσότερο συμμετέχουν οι επενδυτές στις εταιρείες μέσω καλύτερης δυνατότητας συμμετοχή τους στην ψηφοφορία, τόσο καλύτερα θα είναι για μια βιώσιμη ενία αγορά. Εμείς θεωρούμε ότι η καλή διακυβέρνηση θα οδηγήσει σε υψηλότερα κέρδη για τους επενδυτές. Είναι τόσο απλό. Ελπίζω λοιπόν να σας έπεισα ότι ο τρόπος με τον οποίο ε, ε, ψηφίζουμε εξ ονόματος των μετόχων είναι πολύ σοβαρός και αυτή η οδηγία θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας και πιστεύουμε ότι θα έχουν και καλύτερη απόδοση οι επενδυτές μας και θα είναι όλα καλύτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Έχω επίσης και ένα αναλυτικό έγγραφο το οποίο θα σας διανύμω για τα σχόλιά μας επί όλων των διατάξεων της οδηγίας και στη διάθεσή σας για να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο τέταρτος ο μιλητής είναι ο Ζαν Νικολά Καπράς, Διευθυντής της ISS Europe. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την άποψη των πληρεξουσίων συμβούλων. Εγώ θα εκπροσωπήσω την ISS που είναι ένας ε, παγκόσμιος ε, κατεξουδότηση σύμβουλος προς τους θεσμικούς. Βασίζομαι λοιπόν στις ε, πρωτοβουλίες και τις θέσεις που έχουν προωθηθεί τα δύο τελευταία χρόνια. Θα περιοριστώ στο άρθρο 3α, 3α μάλλον, που σχετίζεται με τους πληρεξούσιους συμβούλους, γιατί δεν θεωρούμε σκόπιμο να σταθούμε σε άλλα τμήματα της οδηγίας που σχετίζεται με τους θεσμικούς. Καταρχήν, ποιος είναι ο ρόλος των πληρεξουσίων συμβούλων. Σε υψηλό επίπεδο βοηθούμε τους θεσμικούς επενδυτές να λάβουν τις σωστές αποφάσεις σε σχέση με, με την ψηφοφορία στις γενικές συνελεύσεις. Δηλαδή, όταν ένας πελάτης θέλει να ψηφίσει σε μια γενική συνέλευση, εμείς σε αυτή την περίπτωση του προβάλλουμε μια λεπτομεριακή έκθεση σε σχέση με κάθε ε, σύσταση και πρόταση επιτάπητος. Πολλές φορές εκφέρουμε και αρνητική γνώμη σε συγκεκριμένες ε, προτάσεις ε, διαχείρισης και επίσης αποφαινόμαστε αρνητικά σε σχέση με, την, με τις υπερβολικές αμοιβέ των διευθυνόντων και των υψηλόβαθμων στελεχών. Γι' αυτό ορισμένοι εθνικοί φορείς χρηματιστών προβαίνουν σε συγκεκριμένες δράσεις και λόμπι κατά των πληρεξουσίων συμβούλων. Σε υψηλό επίπεδο υποστηρίζουμε τους ε, τελικούς ε, στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαφάνεια ως προς τη λειτουργία μας. Όμως ε, αμφισβητούμε την αυστηρή ρυθμιστική προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε, το Φεβρουάριο του 2013, λιγότερο από δύο χρόνια πριν, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, η ΕΣΜΑ, υπέβαλε μία προσέγγιση αυτοδιαχείρισης μέσα στα πλαίσια του κώδικα του κώδικα συμπεριφοράς. Και αναφέρω, δεν, έχει, δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με αποτυχία της αγοράς ως προς την διάδραση των ε, πληρεξίων συμβούλων σε σχέση με τους επενδυτές και τους εκδότες. Και γι' αυτό ακριβώς τα συμπεράσματα της ΕΣΜΑ έγιναν μετά από μία ενδελεχή αναθεώρηση του ρόλου των ε, συμβούλων, των κατα... κατεξιοδότηση συμβούλων σε σχέση με την ε, διαβούλευση που γίνεται σε δημόσιο επίπεδο και ε, έγιναν 63 προτάσεις σε σχέση με τους με τους επενδυτές. Πρόκειται δηλαδή για κάτω από 6% των απαντήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. τότε, 6 από αυτούς τους φορείς με τον ISS συμμετείχαν και ο κώδικας συμπεριφοράς δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2014 και οι έξι αυτοί πληρεξούσιοι σύμβουλοι έχουν ε, συμμετάσχει σε μία δήλωση συμμόρφωσης σε σχέση με τις αρχές βέλτιστης ε, πρακτικής. Και όπως γνωρίζετε, η πρώτη αναθεώρηση θα γίνει στις αρχές του 2015. Χρειάζεται λοιπόν τόσο αυστηρή ρύθμιση. Σύμφωνα με την ΕΣΜΑ η απάντηση είναι αρνητική γιατί δεν υπάρχει αδυναμία της αγοράς, η αποτυχία της αγοράς, ούτε υψηλή κίνδυνη. Τι ισχύει σε σχέση με την ανάλυση κόστους ωφελίας και έχετε μπροστά σας τη διαφάνεια. Από πλευρά ευεργετημάτων αμφισβητούμε τα επιπρόσθετα ευεργετήματα που επιτυγχάνονται με την οδηγία γιατί όλες οι προσδοκίες διαφάνειας καλύπτονται από τις αρχές βέλτιστης ε, πρακτικής και επίσης από την δήλωση συμμόρφωσης από πλευράς κόστους η κατάσταση είναι διαφορετική. Όπως ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση οι σύμβουλοι θα επιβαρυνθούν με επιπρόσθετο κόστος συμμόρφωσης, όπως ισχύει με την εφαρμογή της οδηγίας. Σε σχέση με την φύση αυτών των δαπανών, η διαφάνεια ήδη καλύπτεται και αυτό που έχει σημασία είναι ο ρυθμιστικός, η ρυθμιστική μάλλον φύση των προτάσεων. Οι πληρεξούσιοι σύμβουλοι θα πρέπει να ασχοληθούν με τις τρέχουσες δαπάνες εποπτείας διαδρόντας με τους εθνικούς ρυθμιστές. Και αυτό φαίνεται και από την βοήθεια ενός, μιας εξωτερικής νομικής υπηρεσίας που πολλές φορές χρειάζεται. Επίσης, το κόστος εποπτείας θα επιβαρύνει τους συμβόλους, τους συμβόλους με συγχωρείτε, και σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε μεταφορά της οδηγίας στα κράτη-μέλη κατά μη εναρμονισμένο τρόπο. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την τρέχουσα διατύπωση του προσχεδίου οδηγίας, οι σύμβουλοι θα πρέπει να ε, αποκαλύψουν στοιχεία στους ε, πελάτες και στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Εμείς όμως θα πρέπει να αποκαλύψουμε στοιχεία σε σχέση με διαφορές μόνο στους πελάτες και όχι σε άλλους. Αυτό σχετίζεται και με την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, την MIFID, και σε σχέση με τις βασικές υποχρεώσεις πίστεως. Άρα οι οι σύμβουλοι όπως η ISS θα πρέπει να αλλάξουν άρδιν τις επιχειρησιακές δικασίες με βάση το, και το κόστος εποπτείας και συμμόρφωσης. Όπως σας είπα, αυτές οι ταπάνες έχουν υποτιμηθεί ιδιαίτερα σε σχέση με τα στοιχεία που θα πρέπει να ε, αποκαλύψουμε στους εκδότες σε σχέση με την αποτίμηση που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπροσθέτως, φοβόμαστε ότι αυτή, αυτό το επαχθές κόστος συμμόρφωσης θα μπορούσε να έχει ε, επιβλαβείς ακούσιες συνέπειες. Θα αυξήσει το κόστος παροχής υπηρεσιών προς τους θεσμικούς επενδυτές που αντιτίθεται στους ε, βασικούς στόχους της οδηγίας και δεύτερον θα θέσει προσκόμματα και περισσότερη συγκέντρωση και συγκεντρωτισμό στην ίδια τη βιομηχανία, διότι πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε μικρά ε, γραφεία που δεν απασχολούν περισσότερο από 50 εργαζομένους, δηλαδή πρόκειται για ΜΜΕ. Και έτσι χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο για αθέμητο ανταγωνισμό σε σχέση με τους συμβούλους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, οι ίδιοι οι εθνικοί ρυθμιστές θα πρέπει να εποπτεύσουν τις δραστηριότητες μιας πολύ μικρής εταιρεία στη χώρα τους που απασχολεί δύο ή πέντε εργαζόμενους όπως ισχύει στη Σουηδία και την Ιταλία. Επίσης προτείνει να ε, εγγυηθούμε τις συστάσεις των ε, συμβούλων. Πώς μπορεί να υπάρχει εγγύηση εδώ. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα συμβιβασμό δικαιωμάτων σε σχέση με την ελεύθερη διάδοση δεδομένων, δηλαδή ελευθεροστομία των ίδιων των ε, συμβούλων. Και όπως ξέρετε, πουθενά αλλού δεν υπάρχει τόσο υψηλό επίπεδο απαιτήσεων. Συνεπώς, υποστηρίζουμε το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσουμε τη διαφάνεια των πληροεξουσίων σύμβουλων και του τρόπου εργασίας μας, αλλά αυτό ήδη επιτυγχάνεται από τους κανονισμούς που έχει προτείνει η ΕΣΜΑ, όπως ορίζει και ο κλάδος. Επειδή δεν ε, υπάρχει αδυναμία της αγοράς, η αποτυχία της αγοράς θα ήθελα να αναφερθώ στον Γάλλο φιλόσοφο Σάρλ Μοντεσκέ, ο οποίος είπε ότι οι άχρηστοι νόμοι αποδυναμώνουν τους αναγκαίους νόμους. Γι' αυτό εάν υπάρξουν αυστηρά ρυθμιστικά μέτρα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την οδηγία βέλτιστων πρακτικών και σε αυτή την περίπτωση οι σύμβουλοι θα πρέπει να επεξηγήσουν πώς εφαρμόζουν τις αρχές αυτές και να μην υπάρχουν άλλοι επαχθείς όροι για ε, συγκεκριμένες υποχρεώσεις που να τους επιβάλλονται. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Επίσης υπάρχει και ένα γραπτό έγγραφο το οποίο ε, σας επεξηγεί το πώς λειτουργούμε, το οποίο έχει η Γραμματεία της Κριτικής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ήταν Τελευταίος ομιλητής, ο καθηγητής Λούτκαρτ Φαντενμπέρχε, πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής ε, της ΕΚΟΝΤΑ, της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας ε, των Ενώσεων των Διευθυντών, ή κυρία διορθώνουμε, Λούτκαρτ Φαντενμπέρχε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και για την ατότητα μας δίνετε να σας ε, μεταφέρουμε εδώ τη θέση της ΕΚΟΝΤΑ, της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας των Ενώσεων Διευθυντών. Θα ήθελα στο δεκάλεπτο που έχω στη διάθεσή μου Πρώτα απ' όλα να σας ε, αναφέρω τις απόψεις μας σε σχέση με την οδηγία για τους μετόχους, αλλά καταρχάς ε, επιτρέψατε μου κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για την προσοχή που αποδίδεται σε αυτή την πολύ σημαντική συνιστόσα της εταιρικής διακυβέρνησης. Δεν πρέπει να ε, παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι πολλές φορές γίνεται εστίαση, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα διοικητικά συμβούλια. Οι μέτοχοι όμω λαμβάνουν ε, όλο και περισσότερη προσοχή. Επίση συμφωνούμε με τη διάγνωση και τους επιδιωκόμενους στόχους. Ο κ. Κοφεράτη συγκεκριμένα στην εισαγωγική του ομιλία είπε ότι στόχος μας είναι ε, να δρομολογήσουμε εκ νέου την ε, Ευρωπαϊκή Εταιρική Διακυβέρνηση. Πιστεύω ωστόσο Πιστεύω ωστόσο λοιπόν ότι τίθονται και σοβαρά ζητήματα για το κατά πόσον ε, τα διορθωτικά μέτρα που προτείνονται θα φέρουν και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και θα ήθελα να σας ε, εξηγήσω τους λόγους του οποίου δεν συμφωνούμε με αυτά τα μέτρα. Η Οδηγία για τα Δικαιώματα των Μετόχων έχει ως στόχο τη βελτίωση της εταιρική διακυβέρνησης. Το λέει και στην εισαγωγή η Οδηγία. Με εστιάζοντας περισσότερο στα δικαιώματα, ελπίζω βέβαια και στα καθήκοντα των μετόχων ως ε- έλεγκτων της εταιρεία ε, κατά μία έννοια. Η προτινόμενη οδηγία επίσης χρησιμοποιεί ουσιαστικά μετατόπιση της εξουσίας για τη λήψη αποφάσεων, ε, την παίρνει από το Συμβούλιο, το Διοικητικό και εμείς θεωρούμε ότι αυτό σημαίνει έμεση έλλειψη εμπιστοσύνη προ τα διοικητικά συμβούλια. Και επειδή εκπροσωπούμε του διευθυντέ, δεν συμφωνούμε. Το θέμα είναι πώ μπορούν τα διοικητικά συμβούλια να γίνουν πιο αποτελεσματικά όχι να κοιτάμε μόνο τα δικαιώματα των μετόχων. Άρα θα λειτουργήσουν, θα είναι επαρκή τα διαθωτικά μέτρα, διότι, και αυτές είναι βασικές μας παρατηρήσεις, δεν υπάρχει επαρκής κατά την άποψή μας προσοχή στη μεγάλη ανομοιογένεια ε, των μοντέλων ε, μετόχων. Συχνά μιλάμε για θεσμικούς επενδυτές. Σήμερα έχουμε δύο οργανώσεις οι οποίες τους εκπροσωπούν. Όμως δεν είναι η πλειοψηφία αυτών που κατέχουν τι μετοχέ στην Ευρώπη. Και θα έλεγα ακόμη περισσότερο ότι αν δούμε του θεσμικούς επενδυτέ, όπως ασφαλιστικές εταιρείε ή συνταξιδοτικά ταμεία, τα ποσοστά εταιρικών ε, συμμετοχών τους μειώνονται. Από το 28 ε, έπεσαν στο 8% το 2012. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη νομιογένεια. Θα επανέλθω σε αυτό ευθύ αμέσω. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ε, άρουμε τους φραγμούς που υπάρχουν και για το ε, διάσπαρτο μοντέλο και για το μοντέλο ε, που ελέγχουν οι μέτοχοι την κατάσταση. Υπάρχουν προκλήσεις λοιπόν σε ό,τι αφορά το πρώτο μοντέλο, το διάσπαρτο, διάχυτο. Έχουμε ε, αυτή τη μορφή, παραδείγματο χάρη ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ω κανόνα, δεν ισχύει το ίδιο στην υπηρετική Ευρώπη. Πρώτη πρόκληση λοιπόν. Μπορεί αν ενεργεί παθητική μέτοχη να είναι μαζί με του πιο ενεργού και δραστήριου. Ε, είπε και η εκπρόσωπο τη Αβίβα, είπε και η εκπρόσωπο του δικτύου. Βέβαια, η, η ανάγκη είναι να υπάρχει ενδιαφέρον ε, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Υπάρχουν ε, καλές προτάσεις ε, παραδείγματο χάρη να δίνεται περισσότερη προσοχή στα καθήκοντα των μετόχων και την διαφάνεια. Πρέπει όμως να δούμε και άλλα. παραδείγματος χάρη, πώς θα δώσουμε κίνητρα για ενεργό έλεγχο, ε, είναι κάτι που λείπει επίσης ε, το ότι δεν έχουν αρκετά ε, δικαιώματα για τον ορισμό ή την πάυση ενδεχομένως διευθυντών. Και βέβαια θα επιτρέψουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συντονισμένη δράση. Δεν έχουμε βέβαια μόνο το πρόβλημα των παθητικών ή κατακαιρματισμένων μετόχων. Εδώ συζητούμε τα δικαιώματα όχι μόνο στο τέλος του χρόνου, αλλά και για έξι μήνες ε, και τα λοιπά. Τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν όταν λοιπόν περιοριζόμαστε στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο και πώς μπορούμε να διορθώσουμε. Θα πρέπει να έχουμε πιο μακροπρόθεσμους μετόχους, ε, να τους δώσουμε κίνητρα. Βέβαια το επιχειρηματικό μοντέλο των χρηματιστηρίων και των διευθυντών περιοχιακών στοιχείων βασίζεται στις συναλλαγές, όχι στο, στον, ενεργό, στον έλεγχο, στην ενεργή παρακολούθηση. Όσο παραμένει έτσι το μοντέλο θα υπάρχουν προβλήματα ε, για να έχουμε περισσότερο μακροπρόθεσμους και δραστήριους ε, μετόχους. Επίσης χρειάζονται περισσότερες υποχρεώσεις ε, για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και περισσότερη λογοδοσία για τους απληρεξούσιους ε, συμβούλους. Αυτορύθμιση ή υποχρεωτική κανόνες δικαίου. Αυτό είναι μια ε, επιλογή που πρέπει να γίνει. Καλές είναι οι προτάσεις, ε, παραδείγματο χάρη να έχουμε διαφάνεια και για τους θεσμικούς επενδυτές αλλά και για τους ε, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Θέλουμε να είναι πιο υπόλογοι, πιο υπεύθυνοι. Το θέμα είναι τους ε, ελεγκτές ποιος θα τους ελέγχει. Δεν νομίζω ότι ένας συνταξίουχος μπορεί να παρακολουθεί ένα συνταξιοδοτικό ταμείο όπως ε, τις επενδύσεις του. Είναι ένα θέμα λοιπόν είναι κάτι που λείπει αυτό από την οδηγία. Είναι πάρα πολύ ανομοιογενής ο κόσμος, τα συνταξιδοτικά ταμεία, έχουμε ε, τις ε, διάφορες πρακτικές, ε, short selling κτλ. Και δεν έχουμε μόνο καλά παιδιά, δηλαδή αυτούς που ενδιαφέρονται, τους μετός που ενδιαφέρονται και παρακολουθούν ενεργά, υπάρχουν και πολλοί άλλοι πέραν αυτών που έχουν άλλα στο μυαλό του. Δεν θα πρέπει επίση να παραβλέπουν και αυτήν την τέταρτη πρόκληση, το γεγονό ότι υπάρχουν και πολλά άλλα μοντέλα στην Ευρώπη. Πράγματι, σε πολλές χώρες έχουμε ένα άλλο μοντέλο με ε, μετόχους που ελέγχουν κατά κάποιο τρόπο. Και έχει να κάνει αυτό και με σε συνδεδεμένα μέρη. Θα πρέπει όμως να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους μετόχους οι οποίοι ελέγχουν. Μήπως καταχρώνται της εξουσίας αυτής της ελεγκτικής που έχουν. Μήπως θα πρέπει να οριστούν ανεξάρτητοι ε, ελεγκτές. Άρα θα πρέπει να εστιάσουμε και στα δύο μοντέλα και το διάσπατο και το, ε, αυτό των ελεκτών. Πρέπει να είναι επαρκώς ανεξάρτητα διοικητικά συμβούλια. Όχι μόνο στις συνάδειες συνδεδεμένων μέρων. Θα πρέπει να βλέπουμε τη διακυβέρνηση εταιρεία συμμετοχών, αλλά γενικά την ε, εταιρική διακυβέρνηση ε, των ομίλων. Είναι κάτι το οποίο εξετάστηκε και είναι ένα ενδιάμεσο, μεσοπρόθεσμο στόχος ε, στο πλαίσιο του προγράμματος δράση. Αλλά νομίζω ότι την λεγόμενη group governance θα πρέπει να τη δούμε πιο προσεκτικά. Έχουν ληφθεί υπόψη οι συναλλαγέ δεδομένων μερών, τα είπαν οι Ευρωπαίοι εκδότε πριν από εμένα. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω πιο πολύ στο τελευταίο, γιατί η οργάνωσή μα ε, θέλει να είναι αποτελεσματικά τα διοικητικά συμβούλια και νομίζω ότι δεν γνωρίζουμε ε, μάλλον δεν ασχολείται παρκώ με αυτό το στόχο η οδηγία. Δεν θέλουμε μόνο ενεργό έλεγχο ε, και παρακολούθηση από τους ε, μετόχους, αλλά θα πρέπει να είναι σε καλή θέση και οι συμμετέχοντε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και θα πρέπει να εστιάσουμε, περισσότερο την προσοχή μας, γιατί αν στόχος μας είναι οι εταιρείε να εστιάσουν περισσότερο στο μακροπρόθεσμο επίπεδο και οι εταιρείε να εστιάζουν πιο πολύ στην ενεργό παρακολούθηση και έλεγχο σε σχέση με την κοινωνική εταιρική ευθύνη και όχι μόνο ε, στα σφαίρα των μετόχων. Η πτυχή των μετόχων είναι μόνο ένα ε, σκέλο τη όλη διαδικασία παρακολούθηση. και νομίζω ότι η μόνη εγγύηση ε, που μπορούμε να έχουμε ότι δεν θα έχουν ανεγωιστεί όπως θα κοιτάσει τα δικά του συμφέροντα. Η μόνη εγγύηση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει νομικό καθήκον στην Ευρώπη, δηλαδή Μόνο τα εταιρικά συμφέροντα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ε, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι, τέτοιο καθήκον δεν έχουν οι μέτοχοι. Αν κάποιο ασχολείται με το λεγόμενο short selling, μπορεί να μην ενδιαφέρεται ε, αυτός που ασκεί αυτή τη δραστηριότητα για, τη, για το εταιρικό συμφέρον. Επίση, είναι τα διοικητικά συμβούλια οι μόνοι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πού λειτουργεί η επιχείρηση, ποιο είναι το πλαίσιο. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για έλλειψη διαφάνεια σε θέματα ευαίσθητα ε, όταν υπάρχει ζήτημα ανταγωνισμού. Ξέρουν και μπορούν. Και έρχομαι στην καταληκτική μου παρατηρήση. Ποια είναι τα τρία βασικά στοιχεία. Πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο σε επαγγελματίες διευθυντέ, όχι ε, σε δίκτυα ε, φίλων. Και τι δυνατότητες έχουν. Θα πρέπει να αποδείξουν στου μετόχους ότι οι προτάσεις αντιστοιχούν στην ε, στρατηγική. Θα πρέπει να εγγυηθούμε ανεξαρτησία στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και βέβαια σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε και περισσότερα δικαιώματα στους μετόχους αλλά και σε αυτούς ε, ε, της μειοψηφίας, όχι μόνο της πλειοψηφίας. Τελευταίο αίτημα από την πλευρά μας είναι και τα δικαιώματα των μετόχων να είναι προτεραιότητα αλλά και το πώς θα βελτιωθούν τα διοικητικά συμβούλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη σαφή ομιλία σας. Τώρα ερωτήσεις ε, από τα μέλη προς τους ε, διακεκριμένους ομιλητές μας. Έχουμε μια καθυστέρηση ήδη 10-15 λεπτών, οπότε σας παρακαλώ οι ερωτήσεις σας να είναι πραγματικά ερωτήσεις και να είναι σύντομες. Ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, δεν θα ήθελα να είμαι πρώτος, ελπίζω να μην είμαι ο μόνος. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την παραγωγή πλούτου στην Ευρώπη. Όπως μας εξήγησαν οι διάφοροι ομιλητές. Στην τελευταία ομιλήτρια, την κυρία Λούτερ Φαντεμπάγκε, θέλω να της πω ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η ισορροπία που ανέφερε. Τι είναι μια εταιρεία, είναι ένα κεφάλαιο που έχει επενδυθεί, είναι τα διοικητικά στελέχη και είναι και το ανθρώπινο δυναμικό ανθρώπινο δυναμικό, να μην το πω αλλιώ για να μην κατηγορηθώ για μαρξιστής, που συμμετέχουν και αυτοί. Δηλαδή επενδύουν διάφοροι. Επενδύεται ένα ποσό, είναι ένα χρηματοπιστωτικό, μια χρηματοπιστωτική επένδυση. Υπάρχει η γνώση των εργαζομένων και η τέχνογνωσία και υπάρχει και η επένδυση από πλευρά των διοικητικών στελεχών, η τεχνογνωσία η δική του. Και τα ποσοστά ποικίλουν. Κυρία μου, θα θέλατε η νομοθεσία που εξετάζουμε να είναι πιο σαφής μας είπατε. Βεβαίως, μια επιχείρηση χρειάζεται σταθερότητα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι. Χρειάζεται και οι μηχανισμοί, η διαδικασία λειτουργία της να είναι απλές. Αλλά δεν θα ήθελα να καταλήξουμε στο όνομα αυτής της διαφάνειας, ε, σαφήνειας και απλότητας να ξεχνάμε ένα τμήμα αυτών των συμμετεχόντων σε αυτήν την εταιρεία. Ποια είναι η προοπτική σας. Μισό λεπτό. Να συγκεντρώσουμε ορισμένες ερωτήσεις και μετά θα έχετε δυνατότητα να απαντήσετε. Η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή επιλογή εμπειρογνωμόνων κάναμε πολύ ενδιαφέρουσες και σε ένα βαθμό διαφορετικές πρόπτικες για να καταλήξουμε σε μια βέλτιστη σύνθεση. Οπότε, από τους ε, τρεις πρώτους ομιλητές θα ήθελα τη γνώμη τους για την τελευταία παρουσίαση όπου λέγεται ότι τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να είναι πιο ανεξάρτητα, αποτελεσματικά και να λογοδοτούν καλύτερα. Επίσης, άλλη ερώτηση. Τι πιστεύετε για την παρουσία της κυρίας Χέρον, όπου είπατε ότι πρέπει να στηρίζουμε την μακροπρόθεσμη συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών. Θέσατε θέματα λογοδοσίας. Είπατε ότι πρέπει να υπάρχει μία αδιάκοπη αλυσίδα διαφάνειας. Ελπίζω να υπάρξει μία κάποια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των ομιλητών μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο τον λόγο για να θέσει ερωτήσει. Οπότε να δώσω το λόγο στους ε, ειδικού μας να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις που ήδη έχουν τεθεί. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που μου θέσατε. Θίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπου η Γαλλία προηγείται στο πόσο λαμβάνεται υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά έχουμε διάφορα μοντέλα για το πώς να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εταιρική διακυβέρνηση. Εγώ ίδια έχω διαπιστώσει πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση στην Ολλανδία σε σχέση με τη συμμετοχή των εργαζομένων, το Mitbestimmung, στη Γερμανία. Εγώ προτιμώ το Ολλανδικό σύστημα, που είναι αρκετά διαφορετικό από το Ολλανδικό. Οι μεγαλύτερες εταιρείε μπορούν να δώσουν δικαιώματα στους εργαζόμενους, και ιδιαίτερα στους ε, μισθωτούς να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με βάση ορισμένα κοινωνικά κριτήρια. Αλλά οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να είναι εκπρόσωποι των συνδικάτων. Δηλαδή, μία ανεξάρτητη προοπτική, όχι μία μερική προοπτική. Γιατί τότε θα βάζατε στο Διοικητικό Συμβούλιο μία ε, άποψη που εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Για να είναι ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο πρέπει να είναι οι εκπρόσωποι όλων των τμήματων της εταιρεία της, να είναι ανεξάρτητοι. Βεβαίως μπορούμε να έχουμε μια πιο κοινωνική προοπτική και όχι μια καθαρά προοπτική κεφαλαία αγορών. Παρακαλώ εσείς. Κοιτάξτε, θέλω να πω με κάθε σεβασμό, ότι υπάρχουν κάποια λάθη. 49% του ICGN έχουν βάσει στην Ευρώπη. Έχουμε ευρεία ε, εκπροσώπηση. Πρώην πρόεδρός μας ήταν το BlackRock. Αλλά έχουμε και μερικού από του μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές και διαχειριστέ ε, ενεργητικού. Πριν από 22 χρόνια, ο Sir Adrian Cabri, προέδρευσε μιας ε, επιτροπής που έγραψε έναν κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική διακυβέρνηση. Έχει ένα τμήμα που λέγεται τμήμα ε που αναφέρεται στο ρόλο και τις ευθύνες των επενδυτών. Έκτοτε, και μάλιστα ιδιαίτερα μετά το 2010, έχουμε μια σειρά από εθνικά συστήματα. Έχουμε δηλαδή 12 κώδικες δεοντολογίας. Προχωρεί λοιπόν η κατάσταση για το πώς πρέπει να αναλαμβάνουν πιο σοβαρά τις ευθύνες τους οι επενδυτές. Σίγουρα τα διοικητικά συμβούλια έχουν την κύρια ευθύνη για την επιτυχία της εταιρεία. Όταν ε, δημοσιεύσαμε τις ε, αναθεωρημένες, μας, αναθεωρημένες αρχές μας τον Ιούνιο που τις είχαμε εγκρίνει στο Άμστερνταμ, για πρώτη φορά υπήρχε ένα ολόκληρο τμήμα που αναφερόταν στις ε, ευθύνες των επενδυτών. Γιατί αναγνωρίζουμε ότι και οι επενδυτές και τα διοικητικά συμβούλια έχουν συμφέρον να τα πάει καλά η εταιρεία μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω στην ε, ερώτηση για το ρόλο των διοικητικών συμβουλίων. Βεβαίως αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξής μας αλλά κάτι το οποίο ερευνούμε αυτή τη στιγμή είναι οι καταρτήσεις ε, για μη διευθύνοντες συμβούλους. γιατί εκτίθενται περισσότερα σε ε, ζητήματα ε, περιβαλλοντικά και διαχείρισης, άρα θα πρέπει να υπάρχει μία προμπόνο προσέγγιση Γύρω στα 8 χρόνια πριν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ελέγχους, για διαφθορά και ο διευθυντής θα φαινόταν πραγματικά έκπληκτος και δεν θα ήξερε την απαντήσει. Αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις και διευθύνοντας τελέχη που εκπλήσονται και δεν μπορούν να δώσουν μία απάντηση. Γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε την ετήσια γενική συνέλευση για να ορίσουμε τους στόχους. Σε πάση περιπτώσει οι συζητήσεις είναι υψηλότητα του επίπεδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχετε το λόγο. να προσθέσω κάτι σε σχέση με το ρόλο των διοικητικών συμβουλίων. Η Abigail μίλησε για το επίπεδο κατάρτισης, γιατί δεν μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο στο νομοθετικό σκέλος τους κανόνες. Δηλαδή, τα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να χτίσουν το σωστό πλαίσιο λειτουργίας και συμπεριφοράς και αυτό δεν εντάσσεται μόνο στο νομοθετικό πλαίσιο ή αποκλειστικά σε αυτό. Σε σχέση με την οδηγία αυτή λοιπόν, δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει μόνο το νομοθετικό σκέλος, αλλά υποστήριξη για τα διοικητικά συμβούλια γενικότερα. Και δεν νομίζω ότι ζητάμε για καινούριου, δεν μιλάμε για καινούριου κανόνες στην οδηγία καθεαυτή. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε τα θέματα. Ο κύριος Κοφεράτη. Α, με συγχωρείτε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Κοφεράτη, παρακαλώ. Ο κύριος Καβαντά θέλει να πει κάτι. Ε, σας ζητώ συγγνώμη κύριε Κοφεράτη. Θα ήθελα δημοσία να πω στον κύριο Βαντεμπέργκε και σε συναδέλφους της που πολύ σωστά έθεσαν το ζήτημα. Αν είναι η Γαλλία μοντέλο, ε, εγώ δεν το λέω ως ε, Γάλλος, ως Ευρωπαίος μιλάω τώρα. Δεν είναι μοντέλο η Γαλλία και γι' αυτό και με ενδιαφέρει το πώς μπορεί ε, το μοντέλο διοίκησης των μεγάλων επιχείρησεων να βελτιωθεί. Έχουμε τρεις κοπέλους και όχι μόνο στις επιχειρήσεις στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες. Αλλά στη Γερμανία για παράδειγμα που είναι το λιγότερο κακό μοντέλο, για να πω το καλύτερο μοντέλο, ε, είναι καλύτερο. Ποιο είναι το πρώτο, δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα, ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα. Οι επενδυτέ πολλές φορές δεν ελέγχονται ε, καλά στην άσκηση των επενδυτικών του ε, δραστηριοτήτων και πράγματι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το βράχυπρόθεσμο επίπεδο. Υπάρχει διακύμανση Έχουμε 3% μιας διεθνούς εταιρείας εισηγμένης παγκόσμιας ε, ε, τα μερίδια τα πουλάω, φεύγω και ξέρουμε ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό όμως πολλές φορές ε, αποδυναμώνεται ε, το συμφέρον της εταιρείας λόγω αυτή, αυτών των διακοιμάσεων αυτής της ρεστότητας. Θα πρέπει λοιπόν να μην ενθαρρύνουμε ε, αυτές τις βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες ε, στη Γαλλία, έχουμε το ΚΑΚ 40, έχουμε τον Nasdaq, γύρω στις 20 με 25. Αυτές είναι οι πολύ μεγάλες διεθνείς εισηγμένες εταιρείε. Και μέσα σε 30 χρόνια χρηματοοικονομικού καπιταλισμού, με αυτές τις 20-30 μεγάλες εταιρείες, φτάσαμε στην ιδέα, ε, μάλλον οι 20 από αυτές, να είναι σε τουλάχιστον 10 εταιρείε. Δηλαδή υπάρχει ένα είδος ε, πολύ επικίνδυνης συνενοχής ένα κύκλο, σαν διαπλεκόμενα συμφέροντα θα τα χαρακτήριζα. Γιατί δεν υπάρχει πλέον αρκετή ανεξαρτησία. Το είδαμε με την Βιβάντη ε, και με άλλους. Και υπάρχει και ένα τρίτο. ελάττωμα στη Γαλλία. Εγώ ε, διεύθυνα πολλές δημόσιες ε, και ιδιωτικές εταιρείες και είδα ότι Έχουμε και στους συνδικαλιστές πολύ μεγάλη επιρροή από την ιδεολογία για τη δίκηση των επιχειρήσεων. Κατ' εμέ το συνδικαλιστικό κίνημα είναι παροχημένο, δεν έχει προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις και θα ολοκληρώσω με αυτό. Τι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη διοίκηση τελικά. Είναι άνθρωποι που τους, ορίζει, που τους διορίζει το κεφάλαιο, που τους ορίζουν οι επενδυτές και δεν είναι εκεί μόνο για το κεφάλαιο μόνο, αλλά και για την ε, διάρκεια, την ε, διατήρηση και την, ε, τον εξεφρονισμό μιας επιχείρησης. Σε κάποιες γαλλικές επιχειρήσεις δεν τα έχουμε πάει καλά, γι' αυτό και το μοντέλο των γερμανικών οικογενειακών επιχειρήσεων το προτιμώ. Κυρία Βαντεμπέρχη, θα μου επιτρέψετε να επανέλθω στην παρέμβασή σας και σε ό,τι αφορά αυτή την αντίληψη. Αυτό που ήθελα να πω ουσιαστικά Μπορεί να μην τα είπα και πολύ καλά. Όταν μιλάμε για ε, μισθωτό κεφάλαιο, ε, ανέφερα τη Γαλλία ως παράδειγμα γιατί δεν έχουμε το ίδιο παράδειγμα σε πολλές άλλες χώρες. Έπεσε, μιλήσατε για οικογενειακό κεφάλαιο. Ναι, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, αλλά δεν είχα το χρόνο να σας εκθέσω τα πλεονεκτήματα του controlling shareholder αυτών που έχουν δηλαδή τον έχουν ελέγχου μετοχές, αλλά τα οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν είναι ε, ρευστέ ε, και έχουν πρόθεσμο. Αν θέλουμε λοιπόν αυτά τα δύο προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε, δηλαδή αυτή τη ρευστότητα, τη διακύμανση και την έλλειψη ε, ενεργού ελέγχου. Αυτό σίγουρα με τις οικογενειακές επιχειρήσεις δεν υπάρχει ως πρόβλημα. Ευχαριστώ, λέω πρώτος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κοφεράτη για τις καταληκτικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους προσκαλεσμένους μας. Ειλικρινά μας έδωσαν ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Θα επανέλθουμε σε ορισμένα ζητήματα που μας παρουσίασαν και κατά τα τέλη Μαρτίου του επομένου έτους θα ψηφίσουμε μετά από μακρά συζήτηση. Θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα ζητήματα. Εν συντομία. Υπάρχει ένα θέμα που δεν απασχολεί την οδηγία που έφυξε ο κύριος Καβαντά. Δηλαδή, η θέση και το ειδικό βάρος των εργαζομένων. Γι' αυτό η οδηγία θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, δηλαδή της εταιρικής διακυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τους μισθωτούς, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να τους ε, εντάξουμε σε μια εποπτική αρχή. Δεν λαμβάνονται υπόψη από τα διοικητικά συμβούλια, αγνοούνται, ενώ είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο των σφαλμάτων που διαπράττουν οι μέτοχοι και το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή σε σχέση με τη διαχείριση, τη γενικότερη διαχείριση του μετοχικού κεφαλαίου. Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει πολύ μεγάλη σημασία και όλα τα μέσα πληροφόρησης είναι χρήσιμα. Αλλά ε, δεν, ε, δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά μεταξύ του ρόλου που επινοούμε και του έμπρακτου αποτελέσματος. Υπάρχουν διοικητικά συμβούλια που λαμβάνουν αποφάσεις σε σχέση με το CSR, αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ του, ε, αυτού που επινοούμε και του πρακτέου. Βλέπουμε μεγάλες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν εντυπωσιακά έγγραφα για την κοινωνική ευθύνη, αλλά στη συνέχεια χάνουν την αξιοπιστία τους διότι δεν έχουν τηρήσει αυτά τα κοινωνικά συμβόλαια. Οι επιχειρήσεις που δεν είχαν συνεπή στάση σε σχέση με αυτά που προανακοίνωναν και αυτά που πραγμάτωσαν. Δηλαδή υπήρχε διαφορά μεταξύ λόγου και έργου. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα αριθμιστικό πλαίσιο που ορίζει τα δικαιώματα και τους ελέγχους και επαληθεύει τη διαφάνεια. Γιατί δεν πρέπει να μας φοβίζουν ούτε καν οι κυρώσεις. Το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι κυρώσεις έχουν ένα ρόλο αναχέτησης μια συγκεκριμένη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Δεν θα πρέπει να αρκούμαστε σε δηλώσεις βέλτιστης ε, πρακτικής. Θα πρέπει να υπάρξει μία σωστή εξισορρόπηση, χωρίς όμως ε, κανόνες. Δεν σημαίνει ότι η αγορά φτάνει στην ε, θετική αυτορύθμιση. Στην Ευρώπη είδαμε ακριβώς το αντίθετο. Ας φτάσουμε στην καλύτερη εξισορρόπηση και ας δούμε ποια είναι η πραγματική αξία της ρύθμισης και η διάσταση των κυρώσεων. Εάν η Επιτροπή υπέβαλε ένα κείμενο, το έκανε γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι το σχήμα αυτό δεν είναι λειτουργικό και όχι επειδή διαφέρει η κατάσταση από χώρα σε χώρα, αλλά επειδή αυτή η ανισότητα αυξήθηκε ακριβώς λόγω της κρίσης. Και αυτό αφορά τα δικαιώματα όχι μόνο των ε, μισθωτών, αλλά και των ε, μετόχων. Και αν υπάρχει αστάθεια στις αγορές, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουμε κώδικες συμπεριφοράς που δίνουν κίνητρα για καλύτερη συμπεριφορά. Ας εμβαθύνουμε το θέμα της ρύθμισης του κανονιστικού πλαισίου και Ας μην φτάσουμε στο άλλο άκρο της μη ρύθμισης. Καταγράψαμε όλες τις απόψεις, αλλά με απασχολεί το γεγονός ότι ελέγχθη, ότι είναι καλύτερα να μην υπάρχουν ε, και πολλές δεσμεύσεις. Καλύτερα ναι, να μην υπάρχουν δηλαδή δεσμεύσεις και δεσμευτικό πλαίσιο σε σχέση με το αντίπαλο δέος. Εάν κινήθηκε η Επιτροπή προς μία κατεύθυνση, υπάρχει λόγος. Ας το συζητήσουμε λοιπόν. Τι υποκίνησε την Επιτροπή να προβάλλει μια οδηγία σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι σε όλους καλή εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και πάλι τους πέντε εξαίρετους ομιλητές μας που ήρθαν ε, να μας επισκεφθούν. Και ευχαριστώ και όλους όσους ε, παρευρέθησαν σε αυτήν την πολύ σημαντική ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, ε, συνεχίζεται η συνεδρίασή μας. Οπότε, παρακαλώ. Okay, ladies and gentlemen, we can continue our meeting. Συνεχίζουμε παρακαλώ. Thank you for taking... Σας παρακαλώ καθίστε. Λοιπόν, συνεχίζει η συνεδρίαση. Θα περάσουμε το 30. Ανταλλαγή απόψεων για τις ε, μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Δεγκράνδες Πασχουάλ που είναι ο συγητής μας. να θέσω ένα διαδικαστικό. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να συζητήσουμε έχοντας ακούσει πρώτα την Κομισιόν και μετά να ακούσω τους άλλους συναδέλφους και να μιλήσω κι εγώ. Αυτή την διαδικαστική πρόταση θα ήθελα να κάνω. Θα ήταν καλύτερο λοιπόν να μιλήσει η Κομισιόν στην αρχή. ναι, γιατί όχι. Να δώσω το λόγο στην Επιτροπή λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Α, έχουμε και μία παρουσίαση. Λέγομαι Μπαρτόμι Κούτς. Είμαι επικεφαλής της ομάδας για το εταιρικό δίκαιο στην Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Λοιπόν, το πλαίσιο. 98% όλων των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Μόνο 2% έχουν διαμεθοριακή δραστηριότητα. Δηλαδή έχουν θηγατρικές σε άλλες χώρες. Θεωρούμε ότι είναι χαμηλό αυτό το ποσοστό. Υπερβολικά χαμηλό. Υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί. Να έχουμε περισσότερες λοιπόν επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρει η εσωτερική αγορά. Εφόσον θέλουμε ανάπτυξη, απασχόληση, πρέπει να αυξηθεί το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό πνεύμα. Να διευκολύνουμε τους νέους που θέλουν να στήσουν εταιρείες. Διότι, όπως βλέπουμε, δεν τα πάμε και τόσο καλά σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές μας. Είναι χαμηλότερος ο βαθμός δημιουργίας νέων εταιριών έναντι των κυρίων ανταγωνιστών μας. Να διευκολύνουμε λοιπόν πρέπει τη δημιουργία επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων. Να διευκολύνουμε τη δημιουργία τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε, όπου όλα γίνονται επιγραμμικά. Τα συμβόλαια, οι μεταφορές χρημάτων, Τα μητρώα επιχειρήσεων διασυνδέονται και θα λειτουργούν και αυτά επιγραμμικά. Οπότε τι έλεγα, τι έλεγα. Γιατί να μπορούν και να στηθούν οι επιχειρήσεις επιγραμμικά παντού στην Ευρώπη. Έκανε μια συνάντηση με τους πιο επιτυχημένους νέους επιχειρηματίες στην Ευρώπη και τους ρώτησε το εξή απλό τι μπορούμε να κάνουμε για να σας διευκολύνουμε, να διευκολύνουμε την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία. Και μία από τις συστάσεις, συστάσεις τους ήταν να μπορούν να δημιουργούνται στο διαδίκτυο εταιρείε με ενιαία κριτήρια και χαμηλό αρχικό κεφάλαιο για να διευκολύνουμε τη ροή επενδύσεων από τη μια χώρα στην άλλη. Πώς θα το κάνουμε λοιπόν αυτό. έχουμε τη δυνατότητα να μην κάνουμε τίποτα. Να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Αυτό δεν θα βοηθήσει. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε τις προϋποθέσεις για όλες τις ε, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, αλλά αυτό μοιάζει πολύ δύσκολο. Λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές παραδόσεις εταιρικού δικαίου των κρατών μελών. Οπότε, οπότε, θεωρήσαμε ότι ένας τρόπος να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις είναι να προτείνουμε μονοπρόσωπες εταιρείε. Αυτό είναι ο στόχος της πρότασης. Να υλοποιηθεί το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς, να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα, να διευκολύνουμε τη διαμεθοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα, να αυξήσουμε τις επενδύσεις και να ενταχθούμε πλήρως στην ε, ψηφιακή εποχή. Τι προτείνει η πρόταση. Προσφέρει, προτείνει κανόνες για να δημιουργούνται διαμεθορικές επιχειρήσεις. Ένα κοινό όνομα, να υπάρχει ένα ε, ενιαίο μοντέλο για το καταστατικό της εταιρεία, χαμηλό αρχικό κεφάλαιο, κοινοί κανόνες για την προστασία των ε, πιστωτών και κοινή κανόνες διαχείρισης και δυνατότητα να εγγραφούν στο Μητρό επιγραμμικά. Έχουν λοιπόν την επιλογή τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν αυτές τις νέες εταιρείες με όποιο τρόπο θεωρούν πιο πρόσφορο στο νομικό τους πλαίσιο, είτε ως νέα μορφή είτε να την εντάξουν σε κάποια από τις υπάρχουσες. Και αφήνει επιλογή και στους ε, επιχειρηματίες. Αυτή είναι η πιο σημαντική επιλογή. Εάν και κατά πόσο και με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Εάν θέλουν να κάνουν μονοπρόσωπη εταιρεία ή να συστήσουν άλλου είδους εταιρεία εφόσον υπάρχουν αυτές τις δυνατότητες με βάση το εθνικό δίκαιο. Ορίστε λοιπόν, μία συνηθισμένη μικρομεσαία. Υπάρχει μία εταιρεία περιορισμένη ευθύνη, ιδιωτική, σε κάποιο κράτο μέλο και μετά μία θηγατρική σε άλλο κράτο μέλο. Που θα μπορούσε να γίνει με βάση ε, κοινού κανόνε και στα 28 κράτη-μέλη. Λοιπόν, είναι αυτό ευκαιρία ή κίνδυνος. Ακούσαμε πολλά που θεωρούν ότι αυτές οι προτάσεις είναι προτάσεις για να εξισωθούμε όλοι στο χαμηλότερο επίπεδο. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι είναι πρόταση για εξυγχρονισμό. Σε, πολλές, ε, σε πολλά κράτη-μέλη έχουμε απλοποίηση του εταιρικού δικαίου και έχουμε ως ελάχιστο κεφάλαιο ένα ευρώ και απλοποιημένη εγγραφή στα μητρώα εταιριών. Εδώ, στην επόμενη διαφάνεια, βλέπετε ότι σε διάφορα κράτη-μέλη είναι εύκολο να ιδρυθούν αυτές οι εταιρείες αλλά υπάρχουν διάφορες δικλείδες ασφαλείας βέβαια. Αλλά το βασικό είναι ότι το αρχικό κεφάλαιο είναι χαμηλό. Επίσης για την ηλεκτρονική καταχώρηση. Έχουμε ηλεκτρονικά μητρώα και στα 28 κράτη-μέλη και θα διασυνδεθούν. Ήδη έχουμε ένα ηλεκτρονικό πρότυπο μεταφοράς των δεδομένων για τις εταιρείες αυτές, αλλά όχι κατά ανάγκη απευθείας από τον ιδρυτή. Εδώ βλέπετε ότι η επιγραμμική καταχώρηση ιδιαίτερα ε, απευθείας από τον ιδρυτή προς το μητρό είναι δυνατή σε 10. Δεκα... Υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια. Είναι οι χώρες που βλέπετε με κόκκινο. Οι χώρες που ακόμη δεν προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτή η εταιρεία τα αρχικά της λατινικά είναι SUP. Τι προβλέπετε λοιπόν για την εγγραφή της ότι πρέπει να υπάρχουν εθνικοί νόμοι για την ταυτοποίηση και την εξακρίβωση και μπορεί να ιδρυθεί εξ αποστάσεως, επιγραμμικά η εταιρεία χωρίς να ανάγκη κάποιος να πάει κάπου. Τώρα το πώς θα το ρυθμίσει το κάθε κράτος μέλος εξαρτάται από τους ε, κανόνες του κράτους μέλους. Θα πρέπει να υπάρχει μία αρχή Μπορεί να είναι ένας ε, συμβολιογράφος ή ένα σημείο πρόσβασης ή ένας νομικός σύμβουλος που θα αναφέρει τα στοιχεία στην υπεύθυνη αρχή. Το πιο σημαντικό είναι ο ιδρυτής, που είναι ο πιο σημαντικός παράγων, να μπορεί εύκολα και στο διαδίκτυο να ιδρύσει την εταιρεία, όχι κατά ανάγκη από το δικό του κράτος μέλος. Αυτή θα είναι λοιπόν η διαδικασία. Για να συστηθεί μια SUP πρέπει να την γράψετε, θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πρότυπο καταστατικού και θα, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνδεσμος για ε, τα στοιχεία της εταιρείας σε όλα τα κράτη-μέλη. Η εγγραφή αυτή θα γίνει με βάση το εθνικό δίκαιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι με ένα κλικ μπορείς να εγγράφεις την εταιρεία σου σε κάθε κράτος μέλος. Έχουμε 28 διαφορετικές διαδικασίες. Αλλά θα διευκολύνει. Είναι ένα εργαλείο που θα διευκολύνει τη δυνατότητα να ιδρύσει σε άλλο κράτος μέλος μια εταιρεία με απλό τρόπο. Πολλά υπόθηκαν για την ε, έδρα της εταιρείας και ε, τον τόπο εγγραφής. Λοιπόν, θα πρέπει να δεχθούμε ότι μπορεί να υπάρχουν εταιρείε με διαφορετικές έδρες. Οι εταιρείε δηλαδή που ε, εγγράφονται σε μία χώρα ενώ ο ιδρυτής είναι σε άλλη χώρα μπορεί να έχουν διαφορετική έδρα. Και αυτό ισχύει και τις εταιρείε ε, που εξάγουν την ίδρυση μιας άλλης εταιρείας. Επίσης, η συμμετοχή των εργαζομένων και άλλα στοιχεία επαφίενται στις προβλέψεις του εθνικού δικαίου. Τώρα μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, μπορείτε να ρωτήσετε. Ναι, θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει, διότι οι εταιρείε αυτές είναι εταιρείε που θα λειτουργούν με το εθνικό δίκαιο. Γι' αυτό δεν υπάρχουν και αναλυτικές ρυθμίσεις για την ε, μεταφορά της έδρας. Τι θα κάνουμε τώρα για, τις, ε, για τους ψευδώς αυτοαπασχολούμενους ή τις εταιρείε γραμματοκιβώτια. Δεν νομίζουμε ότι αυτό το νομοθέτημα είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτό πρέπει να γίνει αλλού. Νομίζω ότι η σύνδεση δεν είναι επαρκής μεταξύ η συνδεση δεν ειναι μεταξυ αυτων των δύο σε μια σειρά από χώρες μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα, να συστηθεί εύκολα μια εταιρεία, σε άλλες χώρες δεν είναι τόσο εύκολο και το φαινόμενο αυτών των ε, ε, εταιριών γραμματοκιβωτίων δεν σχετίζεται τόσο πολύ με το αν είναι εύκολη ή δύσκολη η ίδρυσή τους. Όμως, εμείς θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε αυτές τις εταιρείες. Δεν θέλουμε αυτές τις εταιρείες, ούτε θέλουμε ψεύτο αυτοαπασχόληση πολύ. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο Κούτσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τώρα ε, θέλει να συνεχίσει ο κύριος Δεγκράντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω θερμά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχε την ε, ευγενή καλοσύνη να προηγηθεί εμού. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ουσιαστικά έκανε, δήλωσε ε, την πίστη του σε αυτό το σχέδιο. Ήταν μια πολιτική δήλωση. Εδώ έχουμε βέβαια κάτι αντίθετο με το χρονικό ενό προαναγγελφέντος ε, θανάτου που ήταν του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος, δηλαδή που το συζητήσαμε χθε. Και άλλους πολιτικούς θανάτους έχουμε βιώσει εδώ που προηγήθηκαν αυτής της εταιρείας ε, SUP. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι ρητή η πολιτική βούληση της Κομισιόν ε, να, να καρποφορήσει αυτό το σημαντικό σχέδιο αυτή τη φορά. Για να μην έχει την τύχη προηγούμενων αυτά τα σχέδια, όπως ε, αυτό που απέτυχε για την Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία, το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας και δεν το ξεχνάμε γιατί πολύ ενθουσιασμό είχε προκαλέσει στην αρχή, υπήρχε συνένεση, τελικά όμως ε, αποσύρθηκε ως πρόταση. Τώρα, σε αυτό το σχέδιο για τη μονοπρόσωπη εταιρεία, πάλι φαίνεται να υπάρχουν οι ίδιοι σκόπελοι με αυτούς που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία. Κάποιες από τις βασικές αρχές του υπερωτικού δικαίου, όπως είναι ο πρώτερος έλεγχος της νομιμότητας, Έχουμε την πειθαρχία κοινωνικού κεφαλαίου για τους ε, πιστωτές, κεντρική διοίκηση, έδρα ή κύρια έδρα ε, ε, εγκατάστασης. Όλα αυτά είναι κάποιοι σκόπελοι. Όμως με καλή πίστη έχει προτείνει αυτά που προτείνει η Κομισιόν και γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συμβιβασμούς γιατί θα πρέπει να έχουμε την ημερική εναρμόνιση και το σεβασμό της επικουρικότητας και πιστεύω έτσι θα φτάσουμε σε ένα επιτυχημένο σχέδιο. Ως εισηγητής τώρα θα ήθελα να, θα έπρεπε ίσως ε, να κάνω έτσι μια πολύ προκαταρκτική εκτίμηση. Ουσιαστικά έχουμε μια πρώτη σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι είναι μια απαραίτητη πρόταση αυτή για τη δημιουργία απασχόλησης ε, και επιχειρήσεων στη εσωτερική αγορά για την ανάπτυξη. Θα τονώσει σίγουρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα έχουμε τον ε, νέο μέτοχο. 6 εκατομμύρια από 20 εκατομμύρια ε, είναι μονοπρόσωπες εταιρείε. Ε, και πράγματι αυτό το βλέπουμε, το είπε και η Κομισιόν, είναι γεγονός. Είναι η τελευταία δυνατότητα να έχουμε ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία ΜΜΕ που θα ευνοεί τη διασυνορική δραστηριότητα, θα μειώνει το κόστος και το διοικητικό άχθος για τη σύσταση εταιριών. Άρα, κατ' εμά χρειάζεται. Χρειάζεται πια προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή. Έχουμε το ψηφιακό θεματολόγιο και ξέρετε ότι είναι προτεραιότητα για την επόμενη πεντέτη, για την Κομισιόν το θέμα αυτό. Έχουμε θετικά επιχειρήματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και διαφορετικά εταιρικά μοντέλα Έχουμε και διαφορετικά συστήματα που εγγυώνται τη σύσταση επιχειρήσεων με μεγάλη ασφάλεια δικαίου. Άρα, ο στόχος είναι να έχουμε αφενός εξυγχρονισμό με νομικά ηχέγγυα αφετέρου. Το άρθρο 14 κατά την άποψή μας και η παράγραφοι 3 και 5 συγκεκριμένα για το μητρό της SUP, θα σας εξηγήσω και στη συνέχεια, μπορεί να είναι μια βάση κάτι τέτοιο. Στην πρώτη αυτή συνάντηση βέβαια που έχουμε, θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των διαφόρων συναδέλφων που πιστεύω έχουν να δώσουν πολλά στην όλη συζήτηση και σας ομολογώ ότι ξεκίνησε επαφές με την κοινωνία των πολιτών και τους άλλους ενδιαφερομένους ε, φορείς. Έχω μεγάλη πολιτική εμπειρία ε, και σίγουρα η εξαποστάσεως ε, νομοθέτηση ε, των αγορών δεν γίνεται. Πρέπει να ακούσουμε τους φορείς επιτόπου, να ακούσουμε τα προβλήματά τους. Να δούμε σε ποιο βαθμό οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνουν και δεν υπονομεύουν ή δεν περιπλέκουν τα πράγματα με νέα μέσα και νομικές πράξεις. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα ε, που μας βρίσκουν σύμφωνος ότι συνιστούν τα εξία και για κάποια άλλα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Είναι επίμαχα, αμφιλεγόμενα. Και νομίζω ότι με την, ε, σε επαφές που θα έχω με την κοινότητα των πολιτών, με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο ε, με τους συναδέλφους, πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα. Το ηλεκτρονικό μητρό είναι ένα θέμα η κεντρική έδρα, κεντρική διοίκηση ή ε, κύρια εγκατάσταση. Νομικές επιφυλάξεις, το ελάχιστο κεφάλαιο που θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα, ε, όπως είναι η απόδειξη φερεγγιότητας ή περιορισμός στην διανομή μερισμάτων, είναι κάποια θέματα. Και τέλος, επειδή ε, δεν μπορώ να τα καλύψω όλα τώρα, είναι η συμμετοχή των εργαζομένων είναι ένα θέμα σημαντικό, τους διοικητικούς υπαλλήλου. και Τέλος, τονίζω ότι πρόκειται για μια οδηγία που δεν επηρεάζει τις μορφές που ισχύουν σήμερα για τη σύσταση μονοπρόσωπων εταιριών περισσότερες σε εθνικό επίπεδο, απλά προσθέτει μια ακόμη ευρωπαϊκή πλέον δυνατότητα, αυτή που λέμε εμείς SUP. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεπάρχουν άλλες μορφές τέτοιων εταιριών. Άρα θα δημιουργηθεί μια νέα εναρμονισμένη μορφή ε, για τα πιο συγκεκριμένα σημεία και θα έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα και αν συνεργαστούμε και έχουμε και την απαραίτητη πολιτική βούληση πιστεύω ότι με βάση την εμπειρία και τα πιο επιτυχημένα μοντέλα θα καταλήξουμε να έχουμε μια ε, νέα μορφή εταιρεία με ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Γιατί στόχος είναι να εγγυηθούμε το καλύτερο δυνατό μοντέλο. Θα επεξεργαστώ λοιπόν τις προτάσεις μου, θα εργαστώ προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα θα είμαι ανοιχτό ε, στις απόψεις ε, και των ομάδων των πολιτικών και των μεμονωμένων λεφτών και στις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών. Απλά η αρχή της διαδικασίας αυτής ήταν σήμερα και τώρα θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Παναλαμβάνω, ε, θα τίνω ευήκον σε όλες αυτές τις απόψεις, ώστε όταν παρουσιάσω την έκθεσή μου να μην ε, είναι στο περιθώριο των απόψεων ε, των ε, συναδέλφων. Αλλά ουσιαστικά να είναι ένα συμπίλημα, μια συγκέντρωση των απόψεων για να έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Regner has the floor. Η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ. Και εγώ προσβλέπω στη συνεργασία και είμαι πεπισμένη ότι η συζήτηση θα προκαλέσει κάποιες ε, καυτές ε, αντιπαραθέσεις. Θα προτιμούσα εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψουμε αυτή την πρόταση. Τα λέω ανοιχτά και να σε εξηγήσω γιατί. Καταρχάς, οι στόχοι της Κομισιόν. Θαυμάσιοι στόχοι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά, είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνουμε τη δημιουργία επιχειρήσεων για να γίνονται με απλό τρόπο. Σαφές. Βεβαίως. Έχουν καλές προθέσεις. Αλλά και οι καλές προθέσεις μπορεί να είναι πλανημένες. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι. Ο στόχος να επιτύχουμε περισσότερη απασχόληση. για να έχουμε και περισσότερη ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντική. Νομίζω ότι είναι κοινικό όμως. Σε χώρες όπου είναι τόσο υψηλή η ανεργία των νέων, να θεωρήσουμε ότι θα δημιουργήσουμε θαυμάσιες θέσεις εργασίας και θα ανθίσει η οικονομία. Γιατί όλοι αυτοί οι άνεργοι νέοι θα γίνουν επιχειρηματίες. Μα δεν υπάρχουν οι συνθήκες αυτές. Θα το επιτύχουμε αυτό όπως είναι τώρα η κατάσταση της, ε, της οικονομίας και δεν θα το επιτύχει αυτό το εταιρικό δίκαιο τους ή άλλους. Νομίζω ότι έχω προβλήματα με την ε, δημιουργία τέτοιων εταιριών. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις το 2012-2013 για το εταιρικό δίκαιο. Βεβαίως αυτά είναι σκόπιμα. Ωστόσο, Θα είχαμε τότε λοιπόν την δυνατότητα με αυτές ε, τις ε, διαβουλεύσεις να ε, συμπεριλάβουμε την κοινωνία των πολιτών. Κάτι έγινε με το διαδίκτυο αλλά δεν ήταν επαρκές. Και αυτό είναι λυπηρό. Διότι η πρόταση αυτή που γίνεται για τη μεταφορά έδρας της Κομισιόν είναι μια καλή δυνατότητα Όμως αυτές οι δυνατότητες για την ιδιωτική ε, ευρωπαϊκή εταιρεία δεν αξιοποιήθηκαν γιατί απορρίφθηκε η πρόταση αυτή από το Συμβούλιο. Αυτά ε, ήθελα να πω καταρχάς και τις επόμενες εβδομάδες θα έχω να πω περισσότερα. Λοιπόν, ε, αυτή η πρόθεση, η κεντρική έδρα να είναι διαφορετική από, την, από τον τόπο της κυρίας εγκατάστασης. Βεβαίως, και εσείς το αναφέρατε, ότι είναι διαφορετικά τα συστήματα στις διάφορες ευρωπαϊκές ε, χώρες για πολύ γνωστούς λόγους και τώρα σε αυτή τη συγκυρία που πάντα θεωρούμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε ε, τη φοροαπάτη έχουμε ε, κάθε λόγο να συμπίπτουν αυτές οι δύο έδρες ούτως ώστε οι εταιρείες να έχουν την έδρα τους εκεί όπου δραστηριοποιούνται και όχι το αντίθετο. Να μην ανοίξουμε την πόρτα λοιπόν σε κάτι άσχημα. Αυτό θα βοηθούσε την εθνική φορολογική νομοθεσία. Και επίσης ε, το δικαίωμα για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση. Δεν αναφέρθηκε. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να φροντίσουμε να πούμε ότι υπάρχει το εθνικό δίκαιο συμμετοχής των εργαζομένων, το οποίο ξέρετε πολλές φορές είναι θεωρητικό, πρέπει να το εξελίξουμε περισσότερο, να το απτύξουμε περισσότερο. Θυμάμαι στην οδηγία για τις υπηρεσίε. επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε παράλληλα δομές που να βοηθήσουν το λεγόμενο φαινόμενο Delaware Έχω πρόβλημα επίσης και με την νομική βάση. Διότι περιορίζεται, μάλλον, συγγνώμη, ε, ο περιορισμός της, του καθορισμού της έδρας σιγά σιγά καταργείται και αντιστρέφεται η κατάσταση. και στην ουσία ε, δίνεται η δυνατότητα να καταστρατηγηθεί το άρθρο 352. Με συγχωρείτε που ε, μακρηγορώ, αλλά υπάρχουν τόσο πολλές επιφυλάξεις για αυτή την πρόταση που είναι σημαντικό να τις αναφέρουμε. Για παράδειγμα, ποιος θα καθορίσει πού μπορεί να προσφύγει κανείς και πώς θα προστατεύσουμε τους πιστωτές, πώς θα προστατεύσουμε τους καταναλωτές από πρώτη άποψη δεν βλέπω τι θα γίνουν αυτά. Έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα. Άρα ποια δικαιοδοσία θα είναι αρμόδια. Ξέρετε όλοι ότι υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η διασύνδεση των μητρώων εταιριών. Έχουμε προπαρασκευάσει αυτή την εργασία. Αλλά αυτή η πρόταση πηγαίνει τόσο μακριά. Γι' αυτό, για να μπορέσει να λειτουργήσει, θα έπρεπε να έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μητρό εταιρεών και δεν το έχουμε. Άρα ο καθένας μπορεί να κρύβεται από τις εθνικές αρχές εάν εγκριθεί ε, η SUP όπως τώρα προτείνεται από την Κομισιόν. Επίσης το αρχικό κεφάλαιο, το ελάχιστο κεφάλαιο, υπόθηκε ότι μπορεί να είναι ένα ευρώ. Και ο εθνικός νομοθέτης δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι εταιρείες θα είναι τρομερός ανταγωνισμός σε αυτά που υπάρχουν. Ε, ε, υπενθυμίζω αυτά που υπόθηκαν για την προστασία των πιστωτών, για την προστασία των καταναλωτών. Όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η πρόταση. Τι άλλο να πω. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Δεν υπάρχουν επαρκείς ε, ε, επίσημες ρυθμίσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ξέπλυμα χρήματος. Και τα συμφέροντα των εμπλεκομένων δεν αναφέρονται ούτε στη διαδικασία ούτε στην πρόταση. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή το συμπέρασμά μου είναι θαυμάσια ιδέα, από πρώτη άποψη, θαυμάσιο, έξυπνο, αλλά άμα το δει κανεί ε, λίγο πιο προσεκτικά, είναι πολύ προβληματικό για τους καταναλωτές, για τους ε, απασχολούμενους, για τους πιστωτές και φυσικά και για τις υπόλοιπες εταιρείες ε, περιορισμένης ευθύνης που ισχύουν με βάση το εθνικό δίκαιο. Οπότε θα υποστούν μεγάλη πίεση αυτές οι άλλες εταιρείες. Ορισμένες ε, είναι μεγάλες εταιρείες. Και θα μπορούσαν και αυτές να δράσουν ως ε, SUP. Σας ευχαριστώ πολύ για το ζωτική σημασία μήνυμά σας, ο κύριος Ράγκεφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς εφαρμόζεται στο εθνικό δίκαιο το εταιρικό δίκαιο και ποια είναι η αξιοπιστία των ξένων εταιριών μεταξύ ε, καταναλωτών και πελατών. Γι' αυτό και οι ΜΜΕ επενδύουν στο εξωτερικό για να μην υπάρχει αυτή η έλλειψη αξιοπιστίας ε, θα αυτοεξαιρεθούν από το καθεστώς των θηγατρικών. και γι' αυτό με αυτή τη μορφή μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ΜΜΕ και να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Η απλοποιημένη διαδικασία ενσωμάτωσης και η ευελιξία αυτού του τύπου της επιχείρησης θα ενθαρρύνουν, θα προωθήσουν την ελεύθερη εγκατάσταση και θα μειώσουν το διοικητικό άχθος μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Επιχειρήν ως προς την επιγραμμική εγγραφή θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, θα πρέπει να ελέγξουμε την προστασία προσωπικών δεδομένων για να μην υπάρχει κακή χρήση των δεδομένων αυτών. Πολλές φορές ε, ίσως ε, το κοινό φτάνει σε λάθος συμπεράσματα. Γιατί μιλάμε για μία μορφή εταιρεία που συνυπάρχει με τις εταιρείε περιορισμένης ευθύνης γενικότερα. Θα πρέπει να υπάρχει η διπλή προστασία των πιστωτών, όπως είπε η Επιτροπή, ελέγχοντας τους ετήσιους λογαριασμούς της επιχείρησης και με μία δήλωση φερεγγιότητας. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μια πιο απλή διαδικασία εγγραφής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ο κύριος που μίλησε από την Επιτροπή να ακούσει την παρέμβασή μου υπό το θέμα 31. Ο κύριος ε, Λεμπρετών. Κύριε Πρόεδρε, αντιτάσσουμε για δύο λόγους ε, σε αυτή την οδηγία για τη δημιουργία της ΣΟΥΠ. Βασιζόμαστε στο άρθρο 50 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ελευθερία εγκατάστασης. Είναι λάθος αυτό. Θα έπρεπε να βασιστούμε στο άρθρο 352 σε σχέση με τις δράσεις που δεν προβλέπονται από το Συμβούλιο, όπου το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφανθεί με ομοφανία. Η νομοθεσία, η απόφαση του 2006 του 10 σχετίζεται με το άρθρο 352 σε μια υπόθεση πολύ κοντά στη δική μας σε σχέση με τη σύσταση επιχειρήσεων. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση ο ενάγων έχασε. Αυτή η νομολογία ισχύει και στη δική μας υπόθεση στο, στα σημεία 40 και 41 των αποφάσεων στοιχειοθετείται αυτό. Μιλάμε για μία ε, ε, μορφή μία δικαιοδοτική μορφή η οποία επικαλύπτει την πρώτη με βάση το άρθρο 352 και εδώ μιλάμε και για, για εθνικό δίκαιο και για συγκέντρωση δεδομένων που αντιτίθενται ε, στο εθνικό δίκαιο. Άρα θα πρέπει να βασιστούμε στο άρθρο 352. Επί της ουσίας η πρόταση έχει πολλά αρνητικά σημεία Νομίζω ότι δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις, υπάρχει ευελιξία, αλλά δυστυχώς υπάρχει μεγάλη ελαφρότητα υπό την αρνητική άποψη του όρου. Οι μονοπρόσωπες εταιρείε και η δημιουργία τους ε, ηλεκτρονικά χωρίς φυσική παρουσία δεν είναι κάτι το σωστό. Υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα. Επίσης η υποχρεωτική εγγραφή μέσα σε τρεις μέρες δεν επιτρέπει στο κράτος τη συναφής παληθεύσεις. Το ελάχιστο κοινωνικό κεφάλαιο του 1 ευρώ είναι γελίο. Ένας και μοναδικός εταίρος επίσης που μπορεί να λάβει αποφάσεις χωρίς γενική συνέλευση είναι κάτι το ανησυχητικό είναι παράλογο να μιλάμε για ενιαίο, ε, ε, για μοναδικό μάλλον ε, εταίρο, είναι οξύμορο σχήμα. Επίσης, η πραγματική έδρα από την καταστατική έδρα επιτρέπει καταχρήσεις. Αυτές οι μονοπρόσωπες εταιρείες στην ουσία δεν θα λογοδοτούν πραγματικά στους πιστωτές και τα κράτη δεν θα έχουν κανέναν έλεγχο στις μονοπρόσωπες, μονοπρόσωπες αυτές εταιρείες. Θα μπορούν να παρακάμψουν το εθνικό δίκαιο ως προς το εταιρικό του σκέλος, θα οδηγήσει στο κοινωνικό ντάμπινγκ και στην ε, διαφθορά καθώς και στη φορολογική απάτη. Η πρόταση αυτή ε, στην ουσία τι κάνει. Υποσκάπτει την εθνική κυριαρχία βασιζόμενη στην αρχή της ε, ε επικουρικότητας. Κυρία Χιουτλάντ. Ευχαριστώ. Πολλά προελέχθησαν από αυτά που θα ήθελα να πω. Συμφωνώ με την κυρία Ρέγνερ και εγώ ανησυχώ για αυτό το πλαίσιο λειτουργίας. Μιλάμε για τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα διασυνοριακά. Γι' αυτό υπάρχει και η Ευρωπαϊκή αυτή αρχή για τη σύσταση εταιριών. Αλλά ε, δεν θα πρέπει να υποσκαπτούν τα ε, συνδικαλιστικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των συνδικάτων. Και δεν υπάρχει ελεύθερη ε, διακίνηση υπό δίκαιους και ίσους όρους. Δημιουργεί κίνητρα για τις επιχειρήσεις να παρακάμψουν τον εθνικό νόμο και το φορολογικό δίκαιο και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να εγγραφούν στα μητρώα ενός κράτους ε, μέλους, ενώ οι βασικές τους υπηρεσίες ε, παρέχονται σε ένα άλλο κράτος. Έτσι μπορούμε να έχουμε ε, επιχειρήσεις γραμματοκιβωτίου, δηλαδή ανύπαρκτες επιχειρήσεις και μπορούν να εγγραφούν ανήκουν σε ένα κράτος το οποίο έχει τη χαμηλότερη φορολόγηση και μισθοδοσία αποφεύγοντας ε, την φορολόγηση στο κράτος όπου πραγματικά λειτουργούν. Έτσι δημιουργείται άδικος και αθέμητος ανταγωνισμός και θα μπορούσαμε να έχουμε μία προς ένα προς τα κάτω ανταγωνισμό σε σχέση με, με τη φορολόγηση και τις συνθήκες εργασίας. Καταλαβαίνετε πού θα μπορούσε να οδηγήσει κάτι τέτοιο. Έτσι δεν υπάρχει δίκαιη μετακίνηση και κοινωνική ευθύνη. Ήδη υπάρχει κοινωνικό dumping σε όλους τους τομείς των κατασκευών της ναυπηγικής, των καινοτομιών και ούτω καθεξής. Και έτσι ρίχνουμε λάδι στη φωτιά προς αυτή την ε, κατάντη προσέγγιση. Έτσι θέλουμε να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Δεν το νομίζω. Νομίζω, όπως είπε και η κυρία Ρέγνερ, θα έχουμε πολύ σκληρές συζητήσεις και ελπίζω να μην είναι αυτό το μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Βιέφκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι που αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ανέφερε όλες μας τις αμφιβολίες ε, για αυτή τη νέα δυνατότητα που ε, προσφέρεται. Κοιτάξτε, είμαστε ακόμη σε φάση οικοδόμησης της ενιαίας αγοράς και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που θα μας επιτρέψουν να υπερβούμε την κρίση που θα μας επιτρέψουν, έλεγα, να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την ανεργία, ιδιαίτερα την ανεργία των νέων. Λυπάμαι, πραγματικά εκφράζω την συμπάθειά μου προς τον εισηγητή μας, τον κύριο Δεγκράντες Πασκουάλ, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα περίπλοκο και ακαθόδες θέμα, και θα πρέπει να βρει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που ήδη ετέθησαν. Ιδιαίτερα τα ερωτήματα που έθεσε η κυρία Ρέγνερ. Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές ε, είναι αιτιολογημένες. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την προσέγγιση που λέει η ε, είμαι κατά, διότι είναι κακή αυτή η πρόταση. Ακούγοντας ε, τους συναδέλφους μου, είχα την εντύπωση ότι θεωρούν ότι τρελάθηκε η Κομισιόν. Πώς είναι δυνατόν να έχει υποβάλει τέτοια τόσο επικίνδυνη πρόταση η Κομισιόν. Αλλά κοιτάξτε, έχουμε πείρα εδώ. Και έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένα ότι η Επιτροπή δεν έχει παλαβώσει. Αν μας έχουν πολλές φορές υποβάλει προτάσεις οι οποίες δεν είναι πλήρεις, οι οποίες δεν έχουν εξετάσει όλες τις επιπτώσεις τους, παρόλα αυτά είναι μια καλή αρχή. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι τροπολογίε θα υποβάλουμε για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Διότι, κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι όπω η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάναμε για το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο. Κάπως έτσι ήταν τότε η κατάσταση. Θυμάμαι την ε, ανταλλαγή απόψεων και μεταξύ των Υπουργών, 27 τότε Υπουργών και την ε, ανταλλαγή απόψεων που είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας. Πρώτα είπαμε όχι, αυτό είναι κακή πρόταση, ούτε θα τη συζητήσουμε. Αλλά κατά την επόμενη και τις μεθεπόμενες συζητήσεις τελικά αποφασίσαμε ότι μπορούσαμε να υποβάλουμε τροπολογίες για να αποκτήσουμε ένα ουσιώδες νέο νομοθέτημα. Φυσικά θα συμμετάσχει και η Κομισιόν η Κομισιόν θα πρέπει να ακούσει τις ερωτήσεις μας, να προσπαθήσει να απαντήσει. Ο εισηγητής δεν θα πρέπει μόνο να εργαστεί με βάση τις πολιτικές του απόψεις, θα πρέπει να επιδιώξει να ακούσει την άποψη και κοινωνικών εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ποιος είναι ο κύριος στόχος μας. Ο κύριος στόχος μας είναι να επιτύχουμε κάτι. Δεν έχει λοιπόν καμία έννοια να πούμε όχι είναι αρνητικό. Αρνητική αυτή η πρόταση. Νομίζω ότι αξίζει να την εξετάσουμε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι τα κράτη-μέλη θα αρχίσουν τώρα αυτόν τον ανταγωνισμό προς τα κάτω. Τα κράτη-μέλη ούτως ή άλλως και τώρα ε, πολλά χρόνια ήδη στην πράξη είναι σε κατάσταση ανταγωνισμού όσον αφορά τις ε, κοινωνικές συνθήκες, ε, τις, τα κίνητρα που δίνουν σε εταιρείε από άλλες χώρες μέλη και σε άτομα από άλλες χώρες μέλη να εργαστούν και να κατασταθούν στη δική τους χώρα. Και αυτό συνεχίζεται. Ναι, μεν ε, ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια αγορά, αλλά στα πλαίσια αυτά κάθε χώρα προσπαθεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τη. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση λοιπόν. Να συζητήσουμε τα θέματα που τίθενται, να συζητήσουμε τους κινδύνους που τίθενται. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ευθύ εξ αρχής ότι όχι το απορρίπτουμε. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση και πρέπει να την δούμε. Ο κύριος ε, Κέστερ. Δεν νομίζω ότι τρελάθηκε η Κομισιόν. Αλλά έχω κάποιες ε, αμφιβολίες για αυτή την πρόταση για αυτές τις μονοπρόσωπες εταιρείες. Βεβαίως θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε απασχόληση, όλοι συμφωνούμε. Αλλά αυτή η πρόταση για τις μονοπρόσωπες εταιρείες βασίζεται σε μια βασική δογματική αντίληψη. Λέμε, δηλαδή, λένε δηλαδή, ότι είναι πολύ αυστηρές οι ρυθμίσεις για την αγορά εργασίας και γι' αυτό πρέπει να μειωθούν οι ρυθμίσεις, να διευκολύνουμε την δημιουργία εταιριών και έτσι θα έχουμε ανάδειξη και απασχόληση. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το βασικό πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη. Επιπλέον, στη Γερμανία έχουμε αρκετή πείρα. Στη Γερμανία είχαμε τη λεγόμενη πολιτική της, του θεματολογίου. Θελήσαμε να μειώσουμε τις... Ε, ε, ρυθμίσεις ε, ε, εργασίας δημιουργήσαμε τις λεγόμενες και εκεί εγώ εταιρείε τις λέγαμε έτσι. Εγώ ανώνυμες εταιρείε. Και αυτή η προσπάθεια απέτυχε πλήρως. Γι' αυτό έχω λοιπόν αντιρρήσεις. Η διευκόλυνση δημιουργίας αυτών των εταιριών δεν θα δημιουργήσει καλές θέσεις εργασίας, μάλλον θα είναι επισφαλεί αυτέ τι θέσει εργασία, θα αυξηθεί η επισφάλεια στην αγορά εργασία. Δεν χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα στην Ευρώπη. Εάν θέλουμε να δώσουμε μια προοπτική εξόδου από την ανεργία για του εργαζόμενου. Κατά λίγο λοιπόν, αυτέ οι μονοπρόσωπε εταιρείε, αυτή η απόπειρα δημιουργεί τον κίνδυνο να υπάρξει ανταγωνισμός προς τα κάτω. Ανταγωνισμός δηλαδή με στόχο να μειωθούν ακόμη περισσότερο ή κοινωνικές προδιαγραφές. Ξέρετε ότι αυτό θα ε, λειτουργήσει πέρα αυτών που αμφισβητούν την Ευρώπη. Και αυτές οι εταιρείε οπωσδήποτε δεν θα επιτρέπουν την συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. Έχω λοιπόν πολλές επιφυλάξεις. Πρέπει να συζητηθούν σε βάθος αυτές οι αντιρρήσεις σε σχέση με τις SUP. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh, Mrs. Ευχαριστούμε κυρία Ρουζιέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, η έκθεση αυτού του σχεδίου προβάλλει στόχους ε, που σίγουρα μας βρίσκουν σύμφωνος. Η ε, ανική εργασία, εύκολη σύσταση εταιριών, αλλά όπως ε, και πολλοί συνάδελφοι, με πρώτη κυρία Ρέγκνερ, έτσι και εγώ, φέτο το ερώτημα μεταξύ αφενός των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας ε, και το στόχο, των στόχων που θα υπηρετήσουν. Θέλουμε και διευκρινήσεις βέβαια. Το θέμα είναι ότι μάλλον δεν είναι η λογική, η λογική της εναρμόνισης ε, υφιστάμενων τύπων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τύπου εταιρείας που έρχεται να προσθεθεί και θα συνεπάρχει με τις ήδη υφιστάμενες μορφές εταιριών. Εγώ πραγματικά ε, έχω κάποιες επιφυλάξεις όταν προσπαθούμε να προσθέσουμε σε ήδη φυστάμενες εθνικές μορφές εταιρεών μια ευρωπαϊκή. Ε, μήπως θα κάνει πιο περίπλοκα τα πράγματα αντί να τα πλουστεύσει και εξηγούμε. Έχουμε οικονομικούς παράγοντες, έχουμε πιστωτές ε, οι οποίοι σε ένα κράτος μέλος έχουν να κάνουν που τις γνωρίζουν καλά το να καταφτάσει τώρα μια πρόσθετη μορφή επιχείρησης, καινούρια, δεν ξέρω σε τι απλούστευση θα οδηγούσε. Ουσιαστικά με αυτό το οριζόντιο ε, μέτρο έχουμε εναρμόνιση χωρίς να το λέμε ξεκάθαρα. Κάθε εθνικό δίκαιο δηλαδή πρέπει ε, τελικά να προτείνει αυτή τη συγκεκριμένη μορφή εταιρεία. Άρα, στο πούμε ξεκάθαρα, πάμε για αναρμόνιση, δημιουργία ενό παράλληλου μέσου εργαλείου. Μάλλον πηγή σύγχυση είναι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Έπειτα, μιλάμε για απλοποίηση, επιγραμμική, ηλεκτρονική σύσταση εταιρεών. Ξέπαινος ο στόχος, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε μια ευρωπαϊκή μονοπρόσωπη εταιρεία να τον πετύχουμε αυτό το στόχο. Θα σας πω τι γίνεται στη Γαλλία ακούμε κριτικές για αυτή τη χώρα, αλλά ίσως πρέπει να δούμε και τι έχει πετύχει, διότι σε ό,τι αφορά τη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, που ενέχει την υποχρέωση εταιρείε που προέρχονται από άλλες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν να εγκατασταθούν σε μια χώρα ή προσωρινά να παράσχουν υπηρεσίες σε ένα άλλο τόπο, σε μια άλλη χώρα προορισμού, θα μπορούν να προσφέρουν ε, στο διαδίκτυο τη δυνατότητα ε, διεκπέρασης αυτών των ε, διατυπώσεων. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά η Γαλλία τι φιλοσοφία επέλεξε. Δεν υπάρχει λόγος, είπαμε, οι επιχειρήσεις από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες από τις γαλλικές επιχειρήσεις. Άρα, έχουμε τη δυνατότητα σύστασης ε, οποιαδήποτε επιχείρησης στο διαδίκτυο, ανεξαρτήτως των τυπώσεων στο, στη Γαλλία και να μπορούν να παρέχουν και υπηρεσίες. Και ανεξαρτήτως δραστηριότητας. Και μάλιστα αυτές και, και για επιχειρήσεις που οι δραστηριότητες δεν εντάσσονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες τώρα η ε, δυνατότητα σύσταση μιας εταιρείας ηλεκτρονικά κτλ. Δεν θα έπρεπε να βασιστούμε στα εφτάμενα εργαλεία και μηχανισμούς και να μην ζητούμε, δημιουργούνται άλλα εργαλεία και έτσι να χάσουμε, να μην είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν θέλουμε να γενικεύσουμε την ηλεκτρονική πρόσβαση, σε επιχειρήσει μια επιχειρήση Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια νέα μορφή ευρωπαϊκής εταιρεία, αλλά να ε, ελαφρύνουμε το βάρος ε, των κρατών και να μεταφέρουμε στο εθνικό δίκαιο τα εφιστάμενα νομοθετήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύσταση αυτού του είδους ε, εταιρείας. Πράγματι, δεν καταλαβαίνω το στόχο. Το είδαμε. Και το τομέα των υπηρεσιών. Ήδη προσφέρονται δυνατότητε στι υφιστάμενε επιχειρήσει να μετεγκατασταθούν σε μια άλλη χώρα, να παρέχουν προσωρινά ε, υπηρεσίε σε μια άλλη χώρα. Στο πλαίσιο όμω τη μεταφορά οδηγία για τι υπηρεσίε του εθνικό δίκαιο, υπάρχουν κάποιε υποχρεώσει ε, για τι χώρε προορισμού και ε, υπήρξαν κάποια θεμητοί λόγοι, προστασία περιβάλλοντος καταναλωτών. Άρα, αφού αυτό είναι ήδη δυνατό σε ποια επιπλέον εναρμόνιση αποσκόπουμε με αυτή τη νέα μορφή εταιρεία. Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος. Εγώ βλέπω εδώ όμως μια νέα απόπειρα να επανέλθουμε στην αρχή της χώρας προέλευσης, της χώρας καταγωγής. Δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε μια εταιρεία που συνιστήνεται υπό τη μορφή αυτής της εταιρεία, οδηγούμαστε σε μεγαλύτερη εναρμόνιση. Ήδη δηλαδή η απλούστευση περιορίζεται. Και γυρίζουμε στην αρχή όπου έχουν το προνόμιο οι χώρες να ορίζουν κάποιες διατάξεις, την προστασία των κοινωνικών, την προστασία του κτλ. Και μια τελευταία εμπειρία που θέλω να σας μεταφέρω για τον τρόπο λειτουργίας ε, της σύσταση επιχειρήσεων στη Γαλλία. Ήδη έχουμε τη δυνατότητα ε, να συστήνουμε μονοπρόσωπες εταιρείε με κεφάλαιο ύψους ενός ευρώ. Είναι ένας μοχλός ε, απλούστευσης, ναι, μεν, αλλά στο, πώς να το πω, για τις υπηρεσίες, την παροχή υπηρεσιών. Το έλεγε και η κυρία Γιούτλαντ. Ήδη έχουμε τη δυνατότητα και για μονοπρόσωπες εταιρείε από άλλα κράτη να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ένα άλλο κράτος. Ανησυχητικό είναι το φαινόμενο που παρατηρούμε σε κάποιους τομείς, δηλαδή να παρακάπτεται η οδηγία για την απασχόληση των εργαζομένων. Το έχουμε συζητήσει πολύ αυτό το θέμα στην προκλητική εκστρατεία. Γιατί ουσιαστικά παρέχει ε, προστασία, είναι μια ασφαλιστική δικλίδα για τους μισθωτούς εργαζομένους, όταν όμως έχουμε αυτοαπασχολούμενους, ανεξάρτητους επαγγελματίε, οι οποίοι έρχονται και ναι, μεν φαίνεται ότι ε, παίρνουν, είναι ανεξάρτητοι μεν, αλλά έχουν τις υπηρεσίες, της ε, συγγνώμη, μισθωτών, ε, τότε παρακάπτεται η απόσπαση με αυτή, η σχετική ε, οδηγία δηλαδή. Όταν δέχονται πιέσεις στα κράτη-μέλη όμως, για να μειώσουν τις κρατικές δαπάνες, και να έχουμε αποτελεσματικό έλεγχο του εργασιακού και κοινωνικού δικαίου είναι κάτι που γίνεται όλο και πιο δύσκολο ως εγχείρημα. Έτσι πρέπει να έχουμε κατά νου αυτή την πτυχή. Και μετά να ξεκινήσουμε με μια μορφή εταιρεία που με το πρόσχημα ε, ότι θέλει να απλουστεύσει τα πράγματα θα δημιουργήσει προβλήματα για το σεβασμό του εργασιακού και κοινωνικού δικαίου στις μέλη. Ευχαριστώ. The, the end of the list of speakers does the... Ο κύριος Ντεγκράντες Πασκουάλ θα ήθελε να λάβει το λόγο. Θα ήθελα να κάνει μια αξιολόγηση η Επιτροπή σε πρώτη φάση και μετά θα λάβω το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να αρχίσω με το γενικότερο μήνυμα που έχει ως εξής. Πολλές ανησυχίες αναφέρθηκαν, αλλά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε να απορριφθεί αυτή η πρόταση. Μπορούμε να επεξεργαστούμε ορισμένα της μέρη για να συμμορφώνεται καλύτερα και να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες ορισμένων ε, μελών του Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ακατόρθωτο να το επιτύχουμε, έτσι ώστε να αρθούν οι επιφυλάξεις. Ως προσφασμένα ζητήματα ίσονος ε, σημασίας, με εξέπληξαν οι παρεμβάσεις ως προς τη νομική βάση γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι βουλευτές θα ήθελαν μια νομική βάση όπου δεν συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Αυτή δηλαδή θα ήταν η κατάλληλη νομική βάση, κάτι το οποίο με εκπλήσει. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που σχετίζονται με το εθνικό εταιρικό δίκαιο και όχι υπερεθνικό. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η νομική βάση είναι σωστή. Σε σχέση με το forum shopping και όλους τους κινδύνους που ελοχεύουν, όπως είπε και ο κύριος Βιέφκα, πολλά συμβαίνουν τώρα και κατά πόσο θα έχουμε μία νέα μορφή εταιρικού δικαίου, αυτό δεν θα αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή αν υπάρχει ένα ενιαίο υπόδειγμα, ένα ενιαίο ελάχιστο κεφάλαιο και ούτω καθεξής, δεν σημαίνει ότι θα δημιουργούνται αναγκαστικά νέες επιχειρήσεις ε, σε σχέση με τις ε, υπηρεσίες μπορούμε να έχουμε συναλλαγές επιγραμμικά μέσω ε, θυγατρικών ή μέσω παροχής υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη. Δηλαδή αυτό είναι συμπληρωματικό η σύσταση εταιρείας. Και πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι ευεργετικό να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες των μονοπρόσωπων εταιριών και αν υπάρχουν παρόμοιοι ομοιόμορφοι όροι σε όλα τα 28 και στα 28 κράτη-μέλη, αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Τώρα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο που είναι γελίο, πολύ χαμηλό, όπως είπε ο κύριος Βιέφκα, δεν τρελάθηκε η Επιτροπή αλλά και τα 16 κράτη-μέλη που προαπαιτούν αυτό το ελάχιστο κεφάλαιο τη στιγμή που αυτό αναφέρεται ως ελάχιστο κεφάλαιο για την εγγραφή. Ισχύει λοιπόν στην πλειοψηφία των κρατών μελών, άρα δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε εφεύρει εμείς. Πρόκειται για μια γενικότερη τάση στα κράτη-μέλη και αυτό περιλαμβάνει και τα μεγάλα κράτη-μέλη. Σε σχέση με τις αμφιβολίες ως προς το ξέπλυμα χρήματος και ούτω καθεξής, νομίζω ότι θα υπάρχει δήλωση φερεγγιότητας και αιτήσιοι λογαριασμοί και ισολογισμός ο οποίος θα ελέγχεται και θα υπάρχουν πραγματικοί δικαιούχοι. Άρα δεν θα υπάρχει ξέπλυμα ως προς τις αρχές εγγραφής. Όπως ξέρετε, έτσι κι αλλιώς αυτές οι αρχές δεν σχετίζονται με θέματα ξεπλήματος και γι' αυτό θα πρέπει να κινηθούμε στην καταπολέμηση της απάτης παρά να τη δημιουργούμε. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούμε να διευθετήσουμε. Θα χαρούμε ιδιαίτερα να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να καταπραϊνθούν αυτοί οι φόβοι. Ναι, Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ την Κομισιόν. Επιμένω γι' αυτό. και για το γεγονό ότι υπερασπίστηκε την πρότασή της. Εγώ ξεκινάω λέγοντας Εγώ νομίζω ότι είμαι πραγματικά θαραλέος που δέχτηκα αυτό το καθήκον. Ξέρω ότι εμείς στην Ισπανία έχουμε αυτή την ε, παράδοση όπως η Ταυρομάχη να δεχόμαστε ε, επικίνδυνες αποστολές. Εγώ είμαι συγητής του Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, πριν πέσω στην πισίνα, κοιτάξω, κοιτάζω αν έχει νερό. Και η Κομισιόν λέει ότι είναι δυνατόν να αποφύγουμε τους ε, σκοπέλους και ότι στόχος μας είναι ακριβώς το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνούμε με την Κομισιόν. Εντάξει, μπορούμε να επιλέξουμε νομική βάση και κάποια νομική βάση που μπορεί να προταθεί μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί η Κομισιόν. Και βλέπουμε ότι ορισμένες προτάσεις που γίνονται μας κάνουν να πιστεύουμε μας κάνουν να φοβόμαστε ότι δεν πιστεύουμε στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι πάντα είναι δυνατόν να συζητήσουμε για την νομική βάση, αλλά να επιλέξουμε νομική βάση που δεν θα δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσει το Κοινοβούλιο, είναι εκπληκτικό. Πρέπει να το συζητήσουμε. Και πρέπει να πούμε εάν συμφωνούμε ή όχι με την πρόταση της Επιτροπής. Ίσως ε, να είναι τελευταία ευκαιρία, γιατί ήδη έχουμε αποτύχει μια φορά. Ίσως να είναι τελευταία μας λοιπόν ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέσο, να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει και αν θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία. Κοιτάξτε, η πραγματική οικονομία και την απασχόληση. Είμαι μια χώρα, όπως ξέρετε, που είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και πολύ ψηλή ανεργία. Αλλά είναι η χώρα όπου αυξάνεται πιο πολύ η ε, απασχόληση. Αλλά βέβαια είναι πολύ σημαντική η ανεργία. Οπωσδήποτε η απασχόληση είναι σίγουρα το πρώτο μας καθήκον. Άρα και εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία γι' αυτό. Στη χώρα μου το 90% της απασχόλησης το δημιουργούν οι μικρομεσαίες, όχι οι μεγάλες. Και ε, βεβαίως χάσαμε τόσε πολλέ θέσει εργασία. Ε, έχουμε 3 εκατομμύρια ανέργου, αλλά δημιουργήσαμε 500.000. Και ε, αυτήν, την απασχόληση δημιουργήσαμε με το νέο νόμο για του επιχειρηματίε. Δημιουργήσαμε νέε προποθέσει για ε, επιχειρηματίε που με την εργασία του και ρισκάροντας τι επενδύσει του τα καταφέρνουν. Είμαστε σε έναν παγκοσμιωμένο κόσμο. Αν η Ευρώπη θέλει να συνεχίσει να είναι ο πρώτος οικονομικός χώρος, δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Διότι ξέρετε υπάρχουν πολλές ε, Και από πολλές ε, πλευρές μας ε, φτάνουν. Λοιπόν, τι κάνει η Κομισιόν. Λέει, θα δούμε αν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ένα νέο μηχανισμό που θα προσπαθήσει να μειώσει τη γραφειοκρατία, τις δυσχέρειες ε, για τη δημιουργία μικρομεσαίων ή και μεγάλων. Μία νέα δυνατότητα που επίσης να προσφέρει και τις ε, εγγυήσει για να μην γίνονται φοραπάτες, για να μην γίνεται ξέπλυμα χρήματος, αλλά να είναι πολύ ευέλικτο μέσο για να δημιουργεί απασχόληση Εντάξει, υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ναι, λίγο. Εντάξει, υπάρχουν και διαφορετικές ιδεολογικές και εθνικέ προσεγγίσεις. Έχουν τεθεί. Και εγώ τι διαπίστωσα κατά την πρώτη εξέταση που έκανα. Τι θέλω να πω λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Ως εισηγητής θέλω να πω ότι θα ακούσω τους πάντες θα εργαστώ, θα λάβω υπόψη της δυσχέρειας και να δούμε εάν θα τα καταφέρουμε να είναι βιώσιμο αυτό το όργανο. Εντάξει, αν τελικά καταλήξουμε ότι είναι αδύνατη αυτή η αποστολή, ε, τότε θα το πούμε. Θα το πω, θαραλέα, με το ίδιο θάρρος που αυτή τη στιγμή την υπερασπίζω αυτή την πρόταση. Ο κύριος Λεμπρετών ήθελε κάτι να προσθέσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για να απαντήσω στην ε, Επιτροπή και τον ε, εισηγητή που ήδη προέτρεξαν ε, εγώ προβαίνω σε μία νομικού τύπου ανάλυση. Δεν θέλω να βραχικυκλώσω το Κοινοβούλιο. Το άρθρο 50 είναι κακή νομική βάση με βάση την απόφαση του δικαστηρίου της Δευτέρας Μαΐου του 2006, αυτό είναι και το έργο μου, να διαβάζω τις αποφάσεις και να τις σχολιάζω. Γι' αυτό είναι εντελώς λανθασμένη βάση το άρθρο 50 καταρχήν. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Αυτά για σήμερα ως προς το σημείο αυτό. Και τώρα θα δούμε τα σημεία 28 και 29 ως προς το πακέτο για το κοινοτικό σήμα. Έχουμε μία έκθεση από την κυρία Βίκστρομ η οποία έχει και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που ξαναγυρίζω στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων σήμερα. Μου έχετε λείψει πολύ όσοι ήσασταν στην προηγούμενη διευθυντή εδώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας ενημερώσω για το πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις για το δεσμετρον για το εμπορικό σήμα. Διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ Κομισιών, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχάς ε, να εκφράσω την ε, ευχαριστίες μου σε όλους τους κοιόδες εισηγητές ε, και τους συνεργάτες, αλλά και στο δικό μου συνεργάτη που κάνει φανταστική δουλειά να ευχαριστήσω και όλο το προσωπικό του Κοινοβουλίου για τις προσπάθειές του. Δεν είναι εύκολο να εργαστεί κανείς ε, για, ε, από την αρχή θα έλεγα, ε, γιατί η παλιά ομάδα που ασχολούμασταν στο το θέμα δεν επανεξελέγησαν ή αποφάσισαν να μην ασχοληθούν με τις ίδιες δραστηριότητες. Να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μου και προς την Ιταλική Προεδρία για τις εξαιρετικές της προσπάθειες. Προσπαθεί να προωθήσει το θέμα παρότι είναι πολύ δύσκολο ενίοτε κάτι τέτοιο. Επίσης ε, και στην Επιτροπή αξίζουν ε, ευχαριστίες γιατί προσπαθεί να εξηγήσει τα πράγματα και να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις προσπαθώντας να εξεύρει συμβεβαστικές προτάσεις. Ε, μια γενική παρατήρηση. Τρεις τριμερείς διαλόγους είχαμε μέχρι τώρα. Πριν από λίγες ώρες ολοκληρώθηκε ο τρίτος τριμερής διάλογος και έπεται ένας τέταρτος για τις 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο συγκεκριμένα. Απα, αναρρύθμιτη ήταν, ήταν και τεχνικές συναντήσεις για να βρούμε λύσεις στα τεχνικά στήματα που δεν έχουμε ακόμη επιλύσει. Επιλύσουμε όμως να τα επιλύσουμε σύντομα. Και είμαι πεπισμένη ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο τελευταία και ότι ακόμη έχουμε τη δυνατότητα να δράξουμε τη στιγμή και να συμφωνήσουμε επί των περισσότερων ίσως των σημαντικότερων ε, πολιτικών συστημάτων που εκκρεμούν. Και αυτό πριν τα Χριστούγεννα. Εάν, και επαναλαμβάνω το εάν, επιδείξουν την απαιτούμενη ευελιξία όλες τις πλευρές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ολοκληρώσει με όλα τα τεχνικά και ή μη πολιτικά ζητήματα. Παραμένουν αποκλήσεις, ε, διαφωνίες που πρέπει να συζητήσουμε και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε και με τους ε, γλωσσομαθείς νομικούς εκ παραλίλου να αναλύουμε τα κείμενα ώστε να είναι τα πάντα συνεκτικά και ξεκάθαρα όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αν συμφωνούν σε κάτι και τα τρία θεσμικά όργανα είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι αρκετά καλό για να διαρκέσει για πολλά χρόνια χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω αναθεώρηση. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να είστε βέβαιοι ότι όλοι εργαζόμαστε πολύ σκληρά και με ως το δυνατό μεγαλύτερη ταχύτητα, χωρίς όμως να υπονομεύουμε την, την ποιότητα του ε, νομοθετήματος. Απλά και μόνο για να ολοκληρώσουμε γρήγορα. Έρχομαι στην ουσία. Με επισημείωση βέβαια, υποσημείωση ότι τίποτα δεν, συμφωνήθηκε πριν συμφωνηθούν τα πάντα γιατί πρόκειται περί πακέτου. Θα επανέλθουμε με το τελικό αποτέλεσμα στην Επιτροπή όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό λοιπόν που προσπαθώ τώρα να κάνω είναι να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση του πώς ε, έχει η κατάσταση με τις διαπραγματεύσεις για να υπάρχει διαφάνεια και για να έχουν οι συνάδελφοι τη δυνατότητα να δώσουν και αυτοί τις απόψεις τους. Πάρα πολλά είναι τα στήματα. Δεν μπορώ να τα καλύψω όλα σήμερα αναλυτικά. Γι' αυτό θα σας παρουσιάσω ποια είναι η βασική μας φιλοσοφία στις διαπραγματεύσεις και εν συνεχεία. Συνοπτικά θα αναφερθώ σε κάποια σημεία που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη. Το Κοινοβούλιο θέλει να εξυγχρονιστεί, να επικαιροποιηθεί ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί σωστά. Θέλουμε το διπλό μοντέλο, το διτό μοντέλο να το προστατεύσουμε, δηλαδή και εθνικά σήματα και σήματα ενωσιακά. Και θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τους χρήστες και από τα δύο αυτά συστήματα. Επίσης, για τη δημιουργία ενός καλού συστήματος για τους χρήστες ε, των εμπορικών σημάτων, αυτό είναι σημείο κλειδί για την διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου. Άρα θέλουμε να κάνουμε κάποια βήματα για εναρμόνιση ορισμένων βέλτιστων πρακτικών στην οδηγία. Σήμερα συμφωνήσαμε επί της αρχής δύο από τα μείζωνα ε, σημεία ε, τριβής, διαφωνίας δηλαδή υποδιαμετακόμιση αγαθά και μικρές αποστολές. Για το πρώτο θέμα συμφωνήσαμε επί της αρχής επαναλαμβάνω ως να δεχθούμε το κείμενο του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα άρθρα. Υπάρχει όμως ε, ε, ανάγκη να κάνουμε κάποιες τεχνικές συζητήσεις. Το Συμβούλιο από την δική του πλευρά δέχτηκε την πρόταση του Συμβουλίου για μια επιπλέον ε, αιτιολογική σκέψη σε ό,τι αφορά τα, τις INN. Ότι δηλαδή τα κοινόχρηστη ονομασίας ε, ε, φάρμακα δεν θα πρέπει να κατάσχονται ε, όταν είσαι διαμετακόμιση σε καμία περίπτωση. Και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε απόλυτα ασφαλές. Για το δεύτερο ζήτημα, τις μικρές αποστολές, θα θέλαμε τα μικρά φορτία Θέλουμε να έχουμε μια διάταξη που θα προστατεύει τα θεμητά συμφέροντα ε, των καταναλωτών, που με καλή πίστη προσπαθούν να αγοράσουν μη παραπημένα προϊόντα. Βέβαια, όσο προσπαθούμε να ε, διορθώσουμε τα πράγματα, τόσο ε, περιπλέκουμε άλλους τομείς. Γι' αυτό στο τέλος συμφώνησε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να απαλείψει ε, από την πρόταση αυτή τη διάταξη για αυτά τα φορτία. Οπότε οι τελωνιακοί θα μπορούν να κατάσχουν παραπημένα πρόταση σε μικρά φορτία χωρίς ε, να καλύπτουν ε, το παράλληλο εμπόριο. Άρα, αν δεν έχει σπάσει κάτι, δεν χρειάζεται να φτιαχτεί. Αυτή είναι η λογική που διέπει αυτή την πρόταση. Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα διακυβέρνηση του οργανισμού που τον γνωρίζετε όλοι ως όχι, το γραφείο δηλαδή για την αρμόνιση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς που είναι αρμόδιο για τα εμπορικά σήματα. Θα έχει μια άλλη ονομασία στο μέλλον και πρέπει να δούμε και τους οικονομικού, τις οικονομικές επιπτώσεις. Νομίζω ότι σήμερα σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο σε διάφορα ζητήματα και παρότι παραμένει ε, άκρος πολύπλοκο το θέμα και δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για όλα τα σημεία, πρέπει να σας πω ότι νιώθω αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε ε, για τα επίμαχα σημεία που απομένουν να έχουμε καταλήξει συμφωνία ίσως και πριν τα Χριστούγεννα. Το Συμβούλιο επέδειξε καλή διάθεση, προθυμία να μετακινηθεί ε, παρότι Έχουμε κάποιες ισχυρές επιφυλάξεις ε, ε, για τη χρηματοδότηση και για τα προτινόμενα μέτρα, διάφορες πτυχές τους, ιδίως για την αντιστάθμιση του κόστους ε, που θα πρέπει να υπομιστούν οι εθνικοί φορείς λόγω του νοσιακού συστήματος. Θέλουμε να είμαστε όμως ρεαλιστές στο Κοινοβούλιο, γι' αυτό θα εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες. Θέλουμε όμως και το Συμβούλιο να δείξει καλή θέληση, εξίσου καλή θέληση σε άλλα ζητήματα για να έχουμε δούνε και λαβίν, αλλά να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Να πω κάποια πράγματα για το άρθρο 12 του κανονισμού και 14 της οδηγίας. Τα άρθρα αυτά καλύπτουν ζητήματα που αφορούν τον δίκαιο ανταγωνισμό και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κατά βάση, τα εμπορικά σήματα δεν θα πρέπει να μπορούν να τα καταχρώνται κάποιοι, για ε, να μην μπορεί να ε, προκαλείται το πλεονέκτημα σε βάρος των ανταγωνιστών. Το Κοινοβούλιο εξετάζει την αρχική του θέση με στόχο μια καλύτερη διατύπωση για να καλυφθούν όλα τα σχετικά ζητήματα ε, τις καλλιτεχνικές εκφράσεις και τα λοιπά, το εξετάζουμε μαζί με εξέχοντες καθηγητές ακαδημαϊκούς από σημαντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ε, με τους οποίους συνεργαστήκαμε πριν από κάποιες ημέρες για το πολύπλοκο αυτό θέμα. Θα σταματήσω σε αυτό το σημείο κύριε Πρόεδρε, όμως ε, θα απαντήσω ευχαρίστως ε, στις ερωτήσεις σας και θα ακούσω βέβαια και τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κυρία Ροζιέρ, ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε ευχαριστώ και για την ίση και την εισηγήτρια για αυτή την πλήρη εισήγηση για την έκβαση των τριμερών διαλόγων. Αυτό που μου τράβηξε την προσοχή είναι τα αγαθά υποδιαμετακόμιση. Πριν από τους τριμερείς διαλόγους είχαμε φτάσει σε μια πολύ καλή θέση με βάση τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που θέλουν να προστατεύσουν την πνευματική του ιδιοκτησία μέσω σημάτων και για την καταπολέμηση της παραχάραξης. Είπατε λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο θα συνταχθεί με το Συμβούλιο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτών θέσεων και οι αποκλήσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση του Κοινοβουλίου και εκείνης του Συμβουλίου. Γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η θέση του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την απάντησή σας. De Grandes Pascual. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Χαίρομαι διότι είχαν πολύ καλή έκβαση τριμερής διάλογου που ήταν τρεις και χαίρομαι εκ των προτέρων για την έκβαση. Ως προς τη χρηματοδότηση φαίνεται ότι βρισκόμαστε στον ε, σωστό δρόμο. Το θέμα αυτό είναι δύσκολο και η ερώτησή μου έχει να κάνει με τη χώρα μου, αλλά εμέσως. Ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Σχολείου του Αλικάντε. Όπως ξέρουμε τα ευρωπαϊκά σχολεία χρηματοδοτούνται από τη ε, εισφορά της Επιτροπής ε, και των κρατών μελών. Σε αυτή την περίπτωση ε, φαίνεται ότι υπάρχει πλεόνασμα, αλλά δεν μπορούμε να αρκεστούμε στο άρθρο 139.3β θα πρέπει να βρούμε μία άλλη βάση για να είναι βιώσιμο αυτό το σχήμα. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει το ζήτημα, αλλά θα ήθελα να μου δώσετε πληροφορίες αν τις έχετε. Ευχαριστώ. Κυρία Βίξτρομ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ προς την άδελφο ε, ε, Ροζιέρ σε σχέση με τα αγαθά υπό διαμετακόμιση. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν κανονισμό για την καταπολέμηση απατών και παραχάραξης. Πρόκειται για την επικαιροποίηση ενός συστήματος. Δηλαδή τα φαρμακευτικά σκευάσματα υπό διαμετακόμιση σε λιμένες ή αερολιμένες δεν θα πρέπει να μην διαμετακομίζονται γιατί αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν. Θα θέλαμε λοιπόν να μην ανασχέσουμε το νόμιμο εμπόριο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για γενώσιμα προϊόντα. που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση. Επίσης, δεν θα πρέπει να ανασχέσουμε οποιοδήποτε νόμιμο εμπόριο. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα στην Επιτροπή αυτή, αλλά στην Ολομέλεια, στην ψηφοφορία Υποβλήθηκαν ε, τροπολογίες που άλλαξαν ε, κάπως την αρχική θέση. Προσπαθούμε να βρούμε λοιπόν ένα συμβιβασμό για να συγκλίνουν οι θέσεις Κοινοβουλίου-Συμβουλίου και δεν απέχουμε πολύ. Αυτό συμβαίνει τώρα. Ξέρετε, όταν διαπραγματευόσαστε, ε, δυστυχώς πρέπει να υποχωρήσετε, να υπαναχωρήσετε και εσείς αλλά και οι άλλοι και πολλές φορές ε, αρκετά. Ως προς τον ε, κύριο Ντεγκράντες Πασκουάλ, ως προς την χρηματοδότηση, το Συμβούλιο ήταν πολύ δημιουργικό, ιδιαίτερα όταν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το τεράστιο πλεόνασμα στην περίπτωση του Αλικάντε. Υπήρξε μια πρόταση για επιπρόσθετους δικαστές, για παράδειγμα ως προς τη χρήση του πλεονάσματος και του σχολείου του Αλικάντε. Εγώ ήμουν εισηγήτρια όταν ασχοληθήκαμε με τη νομική βάση των Ευρωπαϊκών Σχολείων λίγα χρόνια πριν και δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί ένα σχολείο στην Ευρώπη από μία ε, οργάνωση εμπορίου. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, μία διαφορετική αντιμετώπιση των σχολείων. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα ε, σχολείο Mercedes, ένα Volvo και ένα Skoda, δηλαδή ανάλογα από που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησαν να βρουν τρόπους δαπάνης αυτού του πλεονεκτήματος, αλλά δεν έγινε με αυτό τον τρόπο. Μας ενδιαφέρει να μειώσουμε το πλεόνασμα μειώνοντας ε, το κόστος ως προς τα δίδακτρα, για παράδειγμα. Έτσι ώστε οι χρήστες ε, που δημιούργησαν το πλεόνασμα να το χρησιμοποιήσουν. Ελπίζω να φτάσουμε σε μια βιώσιμη λύση και από νομικής πλευράς σωστή. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, Πρόεδρε. Φαίνεται πως όχι. Όχι. Σας ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ για την σαφή ε, παρουσίασή σας της κατάστασης πραγμάτων για το πακέτο για το σήμα. 31 διάφορα. Πρώτον, η Επιτροπή μας θα επισκεφθεί το Λουξεμβούργο αύριο όπου θα ακούσουμε μια παρουσίαση για τις γλωσσικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο. Θα συναντηθούμε με τον ε, Λουξεμβούργιο Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο Υπουργός λέγεται Φέλιξ Μπράζ και θα συζητήσουμε και την επικείμενη Λουξεμβουργέζικη Προεδρία. Επίσης θα έπρεπε η Επιτροπή μας να έχει ψηφίσει για διαπραγματευτική εντολή για τον κανονισμό που απλοποιεί την διαμεθυριακή πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ντελβό. Όμως ε, πρόκειται να γίνει αυτό κατά την επίσκεψή μας, αλλά δεν θα συμμετάσχουν αρκετοί, άρα δεν θα ψηφίσουμε. Επίσης, μας έχει καλέσει σε γεύμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κατόπιν θα συζητήσουμε θέματα όπως η πρόταση αύξησης του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου και στο τέλος, το βράδυ, θα συζητήσουμε στο ελεγκτικό συνέδριο καλύτερες ρυθμιστικές διατάξεις. Ξέρετε ότι ο Κλάους Χάινα Λένε είναι πρώην μέλος της Επιτροπής μας και θα προεδρεύσει σε αυτήν, μάλλον θα είναι ο οικοδεσπότης σε αυτή την τελευταία συνάντηση που θα κάνουμε αύριο. Κάτι άλλο στα διάφορα, οι Επιτροπές Γιούρι και Λίμπε θα διοργανώσουν την ετήσια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου Κατάρτισης ή Δικτύου Δικαστικής Κατάρτισης. Και στα διάφορα ο κύριος Άγνιου έχει ζητήσει επίσης το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω για σοβαρή διαφθορά στο, επίπεδο, στο υψηλότερο επίπεδο των ρωμανικών δικαστηρίων. Μια δική μου εταιρεία που λέγεται Cube Lighting προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε για να εισπράξει ένα χρέος από τη Ρουμανία. Και σε κάθε επίπεδο ε, δικαιοδοσίας των ρουμανικών δικαστηρίων εμποδίστηκε και επιμένω ότι πρέπει επιγόντως να διερευνηθεί το θέμα αυτό. Αυτά που οφείλονται στον ε, ε, ε, πολίτη αυτό από την εκλογική μου περιφέρεια είναι τόσο πολλά που έχασε, έχασαν 16 από τους 34 εργαζόμενους της επιχείρησής τους έχασαν τη δουλειά τους. Μειώθηκε πολύ το, ο κύκλος εργασιών του Όλοι λέμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες. Χρειάζονται λοιπόν, χρειάζεται αυτή η μικρομεσαία τη στήριξή μας και πρέπει να καταλάβουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι το, ε, η διάταξη στα συμβόλαια που υπογράφουν για το ποια δικαιοδοσία, δικαιοδοσία θα ισχύει δεν ισχύει κατά ορισμένε συνθήκε. Και ο δικαστή αρρώστησε την πρώτη μέρα. Ή δικαστή αρρώστησε την πρώτη μέρα τη δίκη. Και τελικά απεδείχθη πω δεν ήταν άρρωστη. Ε, ο άλλο δικαστή που ορίστηκε αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση διότι κατηγορείται ότι δωροδοκήθηκε ακριβώς από το κατηγορούμενο. Έχουν χαθεί διάφορα έγγραφα στραφήκαμε για βοήθεια στην Αλίνα Μπίκα που είναι στο ανώτατο επίπεδο ε, της ε, δικαστικής διαδικασίας αλλά και αυτή πρόσφατα συνελήφθη για λόγους διαφθοράς και στην ουσία υποφέρει ο ψηφοφόρος μου ο ψηφοφόρος της εκλογικής μου περιφέρειας και προσπαθούν προφανώς να τον εξαντλήσουν να εξαντλήσει τις δυνατότητές του και τους πόρους του η λεγόμενη έλεγχοι πριν από την ε, ένταξη μιας χώρας είναι ανεπαρκής αποδεικνύεται και δεν μας εμπνέουν εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτήν την ενημέρωση. Αυτό είναι το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θέλω να σε ενημερώσω ότι αύριο έχουμε αυτήν την εξαιρετική συνεδρίαση της Επιτροπής μας στο Λουξεμβούργο. Η επόμενη τακτική είναι στις 19 Ιανουαρίου 15 μεταξύ 3 και 6.30 και την Τρίτη 20 Πρώτου 15 9 με 12.30 και 3 με, και 3 με 6.30. Οπότε λίγη η συνεδρίαση μα σήμερα. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή και συνεργασία σα.